Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Εξ ονόματος των μελών της ε, Επιτροπής Μεταφορών και των μελών του Κοινοβουλίου και γενικώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαλασορίζω την κυρία Αντινά Βαλεάν. Την καλωσορίζω επίσης τα μέλη της ε, Επιτροπής ΕΝΒΗ. Καλώς ορίζω που θα συμμετάσχουν στην ακροαματική αυτή διαδικασία, όπως και τα μέλη της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Υπό το παράρτημα 6 του εσωτερικού κανονισμού, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μιας κοινή πολιτικής για όλα τα μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα ενιαία έργα όπως ο κοινό, οι κοινοί εθέρες, τα έργα υποδομών, στην ασφάλεια των μεταφορών. Επίσης η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις ε, σχέσεις με τρίτες χώρες και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τους αρμόδιους στα θέματα μεταφορών, όπως και σε σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα υπό τις αερομεταφορές και την αυθυλία της θαλάσσιας μεταφορές, τον IMO. Επίσης, η Επιτροπή Αερομεταφορών παρακολουθεί τις υπηρεσίες ταχυδρομείου και τις τουριστικές υπηρεσίες, και η συνένωση του χαρτοφυλακίου των μεταφορών και του τουρισμού δεν ελήφθη υπόψη και εκφράζουμε την ε, λύπη μας σχετικά με αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κινητικότητα είναι ουσιοδέστατη για τους πολίτες είτε σε αστικό περιβάλλον είτε στο περιβάλλον της υπαίθρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολιτική που θα λειτουργεί προς υπηρεσία όλων των πολιτών και θα ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά στην ψηφιακή οικονομία, στο κλίμα, το περιβάλλον, σε ένα πρότυπο κοινωνικό αποδεκτό από όλους. Η μελλοντική κινητικότητα θα είναι κινητικότητα χαμηλού άνθρακα, προσβάσιμη για όλους, με υψηλή διασυνδεσιμότητα και ασφαλής. Γιατί έχουμε ακόμα 26.000 νεκρούς το χρόνο στις μεταφορές μας. Η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται οπτικά και ακουστικά Χαιρετίζω και καλωσορίζω και όσους μας παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Και διεξάγεται υπό το παράρτημα 7 του ιστορικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει τις δεξιότητες και αρμοδιότητες ως μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων και σύμφωνα με τα καθήκοντα της επιστολής καθηκόντων από την πρόεδρο της Νέας Επιτροπής επί της προσωπικής της ανεξαρτησίας, της δέσμευσης έναντι των πολιτικών που είναι σημαντικές και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της επικοινωνίας. Η Επιτροπή Γιούρια έχει εξετάσει τις ε, χρηματοπιστωτικές καταστάσεις ε, και έχει διαπιστώσει έλλειψη σύγκρουση συμφέροντος. Η κυρία Βαλεάν έχει απαντήσει σε δύο κοινά ερωτήματα υπό την ε, διάσκεψη των Προέδρων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές μεταφράστηκαν σε όλες τις επίσημες γλώσσες και διαναμήθηκαν στα μέλη του Κοινοβουλίου. Πρωτού δώσω το λόγο για 15 λεπτά στην κυρία Βαλεάν θα ήθελα να διαφερνήσω τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε σήμερα. Η κυρία Μελλοντική Επιτρόπος γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία, διότι εσείς οι ίδια είχατε προεδρεύσει σε τέτοιου είδους ακροάσεις. Τα πράγματα λοιπόν θα γίνουν ως εξής. Θα έχουμε την εισαγωγική δήλωση της κυρίας Βαλεάν για 15 λεπτά και όχι περισσότερο. Παρακαλούμε. Θα υποβληθούν 25 ερωτήσεις από τα μέλη. Η σειρά ανά πολιτικές ομάδες και για τους μη εγγεγραμμένους έχει αποφασιστεί από τους πρόεδρους. Ο πρώτος γύρος διανέμεται μεταξύ των πολιτικών ομάδων και στο δεύτερο γύρο έχουν διανεμηθεί ερωτήσεις αναλογικά προς τον αριθμό των μελών. είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε ένα λεπτό να θέσετε την ερώτησή σας. Θα έχει δύο λεπτά απάντησης η κυρία Βαλεάν και μπορεί να τεθεί άμεσα δεύτερη ερώτηση και θα έχετε άλλο ένα λεπτό για αυτήν την δεύτερη ερώτηση. Με απάντηση που δεν θα μπορεί να υπερβεί το ένα λεπτό με τη σειρά της. Αυτές οι δεύτερες συμπληρωματικές ερωτήσεις θα πρέπει να αφορούν, θυμίζω, άμεσα στην απάντηση που θα έχει δώσει ήδη η κυρία Βαλεάν. Θα ζητήσω από όλου να τηρήσουν αυστηρά το χρόνο τους, διότι αλλιώς θα χρειαστεί να σας διακόψω. Το λέω ξανά. Θα έχω την υποχρέωση να σας διακόψω αν υπερβείτε τους χρόνους αυτούς που σας ανέφερα. Έχουμε κάλυψη σήμερα όλων των επισήμων γλωσσών. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε στη μητρική σας γλώσσα προκειμένου να εξασφαλίζετε και η ποιότητα των παρεμβάσεων, να σεβόμαστε και τους διερμηνείς, να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλούμε. Καλό την κυρία Βαλεάν, προτινόμενη Επίτροπο Μεταφορών, να λάβει το λόγο για 15 λεπτά στην εισαγωγική της δήλωση. Παρακαλώ κυρία μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σήμερα κάπως ε, ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε είναι τιμή μου που είμαι υποψήφια επίτροπος ε, για τις μεταφορές και θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου για αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Πρώτα απ' όλα, τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, η ελευθερία να ζήσουν, να εργαστούν και να συναλλαχθούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερω. Αυτό το καθιστά το καθιστούν δυνατό οι μεταφορές, η κινητικότητα και οι μεταφορές συνδέουν έτσι τους ανθρώπους, ενισχύουν την συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση και την ανάπτυξή της. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή καινοτομία και μετασχηματισμού που θα φέρει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα είναι καθήκον μου ως ε, Επίτροπος Μεταφορών να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έτσι ώστε αυτές οι αλλαγές να είναι προς όφελος όλων. Σήμερα ζητάω την έγκρισή σας, την εμπιστοσύνη σας για να κάνουμε τις μεταφορές ε, κατάλληλες για την Ευρώπη, βιώσιμες και δίκαιες. Η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει πει πως το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal θα είναι προτεραιότητα της νέας Κομισιόν. Αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τις μεταφορές. Το Πράσινο Deal θα πρέπει να διασφαλίσει πως οι Ευρωπαίοι θα έχουν μια φθηνή πρόσβαση σε κινητικότητα και μεταφορές. Το δε πρασίνισμα θα πρέπει να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών πρέπει να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομήσει μια συνολική αρχιτεκτονική για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με την ολοκλήρωση του πακέτου καθαρής ενέργειας. Έχουμε τώρα το πιο προχωρημένο πλαίσιο το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε σημαντικές μειώσεις εκπομπών μέχρι το 2030. Αυτό δεν αρκεί. Μέχρι το 2050 θέλουμε να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι και αυτό απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες. Θα εργαστώ σκληρά για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μεταφορών και να συνεισφέρουμε στην ποιότητα του αέρα. Όλα αυτά πρέπει να είναι και οικονομικά επιτυχημένα αν θέλουμε να τα δεχτούν οι πολίτες και να ακολουθήσει ο υπόλοιπο κόσμος. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ε, πολλοί τομείς στους οποίους ε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να αναφερθώ στις ασφαλείς μεταφορές. Σήμερα έχουμε το ασφαλέστερο σύστημα μεταφορών στον κόσμο, αλλά θα πρέπει να το βελτιώνουμε διαρκώς. Η ασφάλεια έχει κορυφαία σημασία για όλα τα μέσα μεταφοράς. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Ασφάλεια από ατυχήματα και από κακόβουλες ενέργειες. Κοιτάζοντας ε, την ε, ασφάλεια, είναι σαφής ο ρόλος των οδικών μεταφορών. Παρά το ότι η Ευρώπη είναι ο ασφαλέστερος χώρος στον κόσμο, 25.000 νεκρή το έτος είναι απλά παράδεκτη. Πρέπει να μειωθούν στο μισό μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2020. Και εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους ε, πόρους ε, σε συνεργασία με υπουργούς και εργολάβους ε, για να το καταφέρουμε αυτό. Μετά, χρειαζόμαστε καθαρή κινητικότητα μέχρι το 2050 σημαίνει ότι θα μειωθούν οι εκπομπές των μεταφορών κατά το 90%. Με τα υφιστάμενα μέτρα όμως θα επιτύχουμε μόνο ένα 20%. Οπότε υπάρχει ανάγκη να κινηθούμε σε τρεις σημαντικούς τομείς. Πρώτον, να δοθούν κίνητρα στις σωστές καταναλωτικές επιλογές, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τρίτον, να αυξηθεί η, και η αγορά καθαρών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η μείωση των αδειών εκπομπών μέχρι καταργήσεως στις αεροπορικές εταιρείες και να επεκταθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών και στην ναυτιλία. Είναι κάτι το οποίο θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή. Γενικά οι χρήστες θα υπομισθούν το κόστος και όχι η κοινωνία γενικώ. Όμως η τιμολόγηση αυτή θα λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες θα είναι διαθέσιμες και προσιτές. Αλλιώς θα έχουμε περιθωριοποίηση ομάδων ή περιοχών, κάτι το οποίο είναι απαραδεκτό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κινητικότητα ως υπηρεσία, να έχουμε εναλλακτικέ στα γεωταχή και να έχουμε έξυπνες συνεργατικές λύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το να περιορίσουμε τις περιτές εκπομπές. Έχουμε παραδείγματος χάρη έλλειψη πρόοδου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αναπτυχθεί επιτέλους αυτό το σύστημα. Αλλά δεν είναι μόνο οι ουρανοί ε, γκριζοί, οι πόλεις υποφέρουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρέπει λοιπόν να μην σπαταλάμε τον χρόνο και το χρήμα των πολιτών. Συνολικά πρέπει να γίνουν όλα τα μέσα μεταφοράς βιώσιμα και γι' αυτό χρειάζεται να βελτιώσουμε όχι μόνο τις προδιαγραφές αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα αναπτυχθούν και θα υιοθετηθούν οι καθαρές λύσεις. Γι' αυτό θα στηρίξω συνεργασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα προστέμενης αξίας. Δεν θα μιλάμε για ε, ανταγωνισμό μεταξύ μεταφορών και κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει αυτά να κινηθούν παράλληλα. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και ιδιώτες επενδυτές ώστε να υπάρξει αύξηση σε σταθμούς ε, φόρτισης ε, και να υιοθετηθούν τα βιώσιμα καύσιμα στις ε, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές για να γίνει ένα μεγάλο άλμα προς την απομάκρυνση από το διοξείδιο του άνθρακα. Μετά θα έχουμε ένα οικοσύστημα έξυπνων μεταφορών πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ψηφιοποίηση έτσι ώστε να γίνουν οι μεταφορές ε, πιο ασφαλείς, ε, πιο καθαρές και πιο πρόσιτες. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι μέρος αυτού του κόσμου, να απολαμβάνουν όλα αυτά τα ωραία της τεχνολογίας και έχουν δικαίωμα. Οι εφαρμογές ε, που αφορούν την κίνηση στα αυτοκίνητά μας και στα άλλα μέσα μεταφοράς. Είναι μερικές μόνο πτυχές που έχουν οι και θα πρέπει να στηρίξουμε την διάδοσή τους. Για τις επιχειρήσεις, ένα περιβάλλον διατροπικών μεταφορών θα τις βοηθήσει να κάνουν οικονομία και να μειώσουν τις εκπομπές. Υπάρχει λοιπόν ένα περιβάλλον ψηφιακών λύσεων και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στην πρώτη γραμμή. Από το blockchain μέχρι την ψηφιακή χαρτογράψη μέχρι τα αυτόματα οχήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία και να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για συνδεδεμένα και αυτόματα μέσα μεταφοράς. Πρόκειται λοιπόν για μια συλλογική προσπάθεια και πιστεύω στην συνεργασία με την βιομηχανία. Αυτό που θα να κάνω και ως πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας και θα συνεχίσω και με τη νέα μου ιδιότητα. Προκλήσεις υπάρχουν, θα επηρεαστούν οι δουλειές. Γι' αυτό θα πρέπει να, δοθούν, να γίνουν επενδύσεις ε, στην επανακατάρτιση των ανθρώπων. Έρχομαι τώρα λοιπόν στην κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Για τους εργαζόμενους στον κλάδο θέλω να εκπαιδευτούν ε, και να επανεκπαιδευτούν αυτοί οι οποίοι κάνουν το σύστημα να λειτουργεί σήμερα. Η αυτοματοποίηση θα φέρει μεγάλες αλλαγές, αλλά ε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το πληρώσει το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης. 11 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν σε αυτό τον κλάδο και δεν θα τους απογοητεύσουμε. Θα υποστηρίξω ένα πακέτο δίκαιης μετάβασης. Οι δουλειές αυτές πρέπει να είναι ελκυστικές για όλους, ειδικά τους νέους, τους οποίους πρέπει να προσελκύσουμε στον κλάδο. Επίσης υπάρχει η πλατφόρμα γυναίκες στις μεταφορές ε, και θα ήθελα να δω την δυνατότητα ισορροπίας ε, των φύλων. Πρόκειται για ένα δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης ανεξαρτήτως ειδικών αναγκών ή εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι πολίτες να κινούνται όλοι σε απομακρυσμένες περιοχές να συνδεθούν και όλοι βεβαίως αναμένουν να προστατεύονται. Η Ευρώπη θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσει ένα τέτοιο συνοπτικό πλαίσιο σε δύο αφορά τα θέματα αυτά για να προχωρήσουν. Τώρα, μιλάμε για τις επενδύσεις, γιατί για όλα τα προγράμματα που χρειάζεται φυσικά η σωστή χρηματοδότηση. Και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο προπολογισμό το 2020 είναι πολύ σημαντικό γιατί αποτελεί μια γέφυρα για το επόμενο πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι απαραίτητο για τη συνέχεια των εργών. Το Connecting Europe Facility θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο πολύτιμες ε, συμβολές μας ως ε, βουλευτές εδώ. Με τον Ντομινίκ Ρικέ συνεργάστηκα για να πετύχουμε να μπουν τα στοιχεία αυτά τα οποία αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για την χρηματοδότηση στις μεταφορές για το κεντρικό δικτυό μας. Ε, μας λείπουν ακόμα βασικοί σύνδεσμοι για τις ε, κοινότητές μας. Δεσμεύομαι ότι θα προασπιστώ τον ε, προπολογισμό για το Connecting Euro για την επόμενη πολιτεστημονικό πλαίσιο. Οι υποδομέ ε, για τι μεταφορέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ για το μέλλον τη Ευρώπη και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι βελτιωμένη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τι υποδομέ και επίση ε, τι ε, εγκαταστάσει διτή χρήση βασική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν καθολικά. Και η υποψήφια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη ότι σε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παγκόσμιο προσκήνιο, ω παγκόσμιο παράγοντα. Θα πρέπει η Ευρώπη λοιπόν να αποτελεί κόμπο για όλε τι γειτονικέ περιοχέ, αλλά και για τι παγκόσμιε ε, αλυσίδε προμήθεια και τι ροέ πελατών. Αυτό χρειάζεται για τον ανταγωνισμό μας, για την ανταγωνιστικότητά μας. Στις μεταφορές λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη ρυθμιστικό μας πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να καταστεί το πρότυπο για όλα τα θέματα. Σε διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τον, ε, τον ΠΟΕΚ θα πρέπει να προωθήσουμε και τις δική μας ε, επιτυχίες για τον ανταγωνισμό, για το περιβάλλον, για την ασφάλεια και το καθεξής. Κυρίες και κύριοι, η εξισορρόπηση των φιλόδοξων ε, οραμάτων για την ε, αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, για τη βιωσιμότητα, με τις αναπτυσσόμενες ανάγκες για την κινητικότητα, για μια ίση και σωστή μετακίνηση με τον ανταγωνισμό θα αποτελέσουν όλα αυτά προκλήσεις μεγάλες για όλους μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι, μιας και σημαντικό είναι μάλλον να υπάρχει συνεργασία με τον ε, με την Επιτροπή και να χρησιμοποιήσουμε την ε, τεχνογνωσία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν δεσμεύομαι ότι εξ αρχής θα συζητάω μαζί σας τις ιδέες για τα διάφορα έργα και θα συζητάμε μαζί την επικείμενη νομοθεσία. Ζητώ λοιπόν την υποστήριξή σας σήμερα προκειμένου να ξεκινήσουμε από μαζί αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Merci Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δήλωσή σας, την παρουσίασή σας και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πάρα αυτά με τον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Το λόγο έχει ο Σβέν Σούλτσε, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία συνάδελφε Βάλεαν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη αυτή εντύπωση που μας δίνεται σε σχέση με αυτά που θα παρουσιάσετε τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Ε, το χαρτοφυλάκι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλές νομοθετικές δυνατότητες διαμόρφωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι είστε συνάδελφος εδώ και πολλά χρόνια, από το 2007 είστε μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως ξέρετε και στην προηγούμενη θετία πολλά πράγματα ήταν ε, αυτά που δρομολογήθηκαν ακόμα και κάποια Και η Ουρσουλα von το ανέφερε, έβαλε στο επίκεντρο την ε, νέα αυτή πράσινη συμφωνία, New Green Deal, και δήλωσε ότι στο σημείο αυτό θέλει να δρομολογήσει γρήγορα αλλαγές. Και εδώ θα συμμετέχει και ο τομέας των μεταφορών στο New Green Deal. Κινητικότητα, λοιπόν, θα πρέπει να την αντιληφθούμε ως υπηρεσία είναι σημαντική αυτή η αλλαγή και έτσι οι υπηρεσίε κινητικότητα θα μπορούσαν να διδεχθούνται από διάφορου παρόχου. Αν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ε, πολύπλευρη παροχή υπηρεσιών, ε, είναι σημαντικό. Ένα παράδειγμα είναι το ΕΛΣΕΚ. Είναι τώρα θα κάνω την ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι νομοθετικές προτάσεις έχετε υπόψη να κάνετε για τον τομέα αυτό προκειμένου να υπάρχει μια συμβολή προς την ε, πράσινη αυτή νέα συμφωνία. Η κυρία Βαλέαν, λέει πρόεδρο, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Η πρώτη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχουμε ουσιαστικά μπροστά μας. Εδώ θα κάνω κάποια γενικά σχόλια. καταρχά, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα επισέλθουμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειε. Χρειαζόμαστε όμω τα πάντα σε αυτή την πράσινη συμφωνία. Και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι έχουμε μια ολική προσέγγιση στην παρούσα φάση. Χρειάζονται λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και όλοι θα πρέπει να συμμετοχούν. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματο, θα πρέπει να αναπτύξουμε βιώσιμε λύσει και να μειώσουμε το αποτύπωμα του με των μεταφορών. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι οικολογικά βιώσιμα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συνολική προσέγγιση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να πετύχουμε. Αν ξεκινήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε αυτά τμηματικά και μόνο, χωρίς συνολική προσέγγιση, η προσπάθεια δεν θα αποφέρει τους καρπούς που ελπίζουμε. Κύριε Σούλτσα, στην κινητικότητα ως υπηρεσία, ως ε, τμήμα του μέλλοντος μας. Η κινητικότητα ως υπηρεσία ακούγεται πολύ θετική. Φυσικά θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η κινητικότητα ως υπηρεσία και από εκεί και πέρα να αναπτύξουμε την ιδέα αυτή. Ακούμε διάφορες ιδέες, ε, διάφορες προτάσεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να εξετάσουμε ακριβώς το χρονικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορούμε να θέσουμε για να μπορέσει η κινητικότητα να αποτελέσει υπηρεσία με πολυτροπικό τρόπο, όπως είπατε, γιατί αυτό είναι απαραίτητο στο νέο αυτό Green Deal, στην νέα Πράσινη Σύμφωνια. Αν θέλουμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα, λοιπόν, θα πρέπει πάνω απ' όλα να επενδύσουμε σε πολυτροπικές μεταφορές. Αυτό πραγματικά είναι κρίσιμη σημασία. Σε ευχαριστώ. Κύριε Σούλτσα, έχετε πάλι το λόγο για την επερώτηση. Και Μία διευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Έχω υπόψη μου την Ήπεθρο, που είναι πολύ αραιοί παρακατοικημένες οι περιοχές αυτές, σε ένα μοθετικό πλαίσιο. Έχετε σκοπό και εκεί να κάνετε προτάσεις ό,τι αφορά τις υποδομές και την κινητικότητα. Κύριε Βαλέα, να απαντήσετε. πατά το κουμπί κάθε φορά γρήγορα γρήγορα. Οι απόμακρε περιοχές είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τις μεταφορές, γιατί εκεί ο κόσμος και η ζωή του εξαρτάται από την διασύνδεση που υπάρχει. Είναι άρα ύψη της σημασίας. Αυτές οι περιοχές ε, με δύσκολη πρόσβαση. Οι απομακρυσμένε περιοχές εκεί θα πρέπει να αναπτύξουμε και να ολοκληρώσουμε το κεντρικό δίκτυο, να υποστηρίξουμε το ρόλο των λιμένων και των αερολιμένων σε τέτοιες ε, περιοχές και προφανώς αυτό ακολουθώντας τους κανόνες του ανταγωνισμού. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άλλη επικάλυψη σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Όταν δεν υπάρχει επαρκή χρήση τουλάχιστον. Αλλά όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τα έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί προκειμένου να διασυνδεθούν Αυτέ οι περιοχές ε, θα χρειαστούν προσπάθειες και αυτό είναι δικαίωμα των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνιελσον για δύο λεπτά. Όχι, ένα λεπτό. Στο συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την οριστή ε, επίτροπο για την εισαγωγή τη. Ε, κάτι που ίσως δεν τονίζεται αρκετά στην επιστολή καθηκόντων αλλά και Στι απαντήσει που μα αποστείλετε είναι οι συνθήκε εργασία αυτών που εργάζονται στον κλάδο των μεταφορών. Σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι μεταφορών εξαναγκάζονται σε ανταγωνισμό ο ένα με τον άλλον ω προ συνθήκε εργασία του και του μισθού του. Αυτό είναι απαράδεκτο επί τη αρχή, αλλά υποσκάπτει και τον ίδιο το τομέα. Έχουμε πρόβλημα προσέλκυσης εργαζομένων στον τομέα αυτών. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών οι καλές συνθήκε εργασία είναι κλειδί για το μέλλον του συστήματος μεταφορών. Επομένως, ως αρμόδια επίτροπο για τις μεταφορές, τι πολιτικές θα ακολουθήσετε προκειμένου να βελτιώσετε τις συνθήκε εργασία στον κλάδο αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντάνιελσον για την ερώτησή σας. Στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ανέφερα σύντομα, γιατί δεν είχα χώρο επέκτασης, αν θέλετε, χρονικά, ότι προκειμένου να επιτύχουμε με οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη των πολιτών. Γιατί οι μεταφορές στους πολίτες απευθύνονται και τους πολίτες αφορούν. Έχουμε τους εργαζόμενους στον τομέα αυτών και έχουμε και τους χρήστες. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες τους και των μεν και των δε, διότι αλλιώς δημιουργούνται κοινωνικές εντάσεις. Μιλώντας για τις συνθήκες εργασίας στον κράτο των μεταφορών, γνωρίζω ότι υπάρχουν ελλείψεις Γνωρίζω ότι υπάρχει ανησυχία σχετικά με την αυτοματοποίηση του μέλλοντος ή την ψηφιοποίηση και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός να βρούμε την κατάλληλη πολιτική ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο για την επανακατάρτιση και τη χρηματοδότηση αυτής της επανακατάρτισης των ανθρώπων αυτών και να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι το μελλοντικό, ότι το μέλλον μάλλον των μεταφορών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα μείνει πίσω. Θα παρακολουθήσουμε εξάλλου και όλη την προσπάθεια στο πεδίο αυτό. Γνωρίζω ότι η προηγούμενη Επιτροπή επ' αυτού εργαζόταν και το Κοινοβούλιο εξάλλου. Είμαι βέβαιο ότι από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε κάτι από το για τους εργαζόμενους. Thank Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ντάνιελσον, ε, για την απάντηση. Θα σας ζητούσα όμως να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και αναφέραμε στις αερομεταφορές πιο συγκεκριμένα εγώ. Η ίδια η Επιτροπή έχει καθορίσει διάφορες πρακτικές που είναι αμφίβολες και που στρεβλώνουν και τον ανταγωνισμό στον τομέα των αερομεταφορών. Επομένως, ε, πιο συγκεκριμένα, πώς θα εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις ε, παρούσες κοινωνικές και εργασιακές διατάξεις στις αερομεταφορές, αλλά εξίσου σημαντικό, θα υποβάλλετε νέα πρόταση νομοθεσίας για τις κοινωνικές συνθήκες στις αερομεταφορές, ως μέρος ευρύτερης δέσμης για τις αερομεταφορές. Επίσης, για παραπλανητικές έδρες ή πλαστά κοινωνικά πιστοποιητικά, ώρες πτήσεις και τα λοιπά και διάφορες πρακτικές που σήμερα σημειώνονται σε αερομεταφορές και είναι κακές, πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Ο τομέας των αερομεταφορών, λέει η κυρία Βαλεάν, είναι εξαιρετικά σημαντικός για το σύστημα των μεταφορών, εξαιρετικά σημαντικός για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες στην Ευρώπη. Οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα αυτών είναι υψηλής εξειδίκευσης. Υπάρχουν όμως αθέμητες πρακτικές όπως είπατε, πράγματι, και συνθήκες εργασίας κακές που δίδουν μια κακή εικόνα στον τομέα. Και εδώ αντιμετωπίζουμε έλλειψη και υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω του κόστους εργασίας των πιλότων, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας που μπορεί να οδηγεί ή να διευκολύνει, αν θέλετε, αθέμητες πρακτικές και πρότυπα επιχειρηματικότητας, χρειαζόμαστε να συμμετάσχουν όλοι οι αερομεταφορείς, οι ενώσεις των εργαζομένων και των εταιριών και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο αν καταβληθεί κοινή προσπάθεια. Ε, πρέπει να, να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος, κυρία μου. Ναι, ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Ε, ήθελα απλώ να πω ότι θα λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο νομοθετικό ή μη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ε, ελλείψεις στα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάουθα Ντίαθ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Θα μιλήσω στα Ισπανικά, πρόεδρε. Κύριε, κυρία, με συγχωρείτε, οριστήσα επίτροπος, ε, οι επιβάτες στις ε, αερομεταφορές το 2018 ε, υπέφεραν 19 εκατομμύρια ε, λεπτά καθυστέρησης. Επίσης υπήρχαν πολλά χιλιόμετρα παραπάνω εκτροπών των πτήσεων. Το 60% των καθυστερήσεων προκαλούνται στην ε, ε, υπερχρησιμοποίηση των αεροδιαδρόμων, ε, το οποίο είναι σημαντικό πρόβλημα για τις αερομεταφορές. Ένα πιο καλά οργανωμένο σύστημα στους εθέρες θα σήμαινε ότι θα είχαμε και πολλά εκατομμύρια λιγότερους τόνους διοξιδίου του άνθρακα ως εκπομπές από τον τομέα συνολικά. Εσείς λοιπόν θα είστε η Επίτροπος που επιτέλους θα ολοκληρώσει τον κοινό ευρωπαϊκό ουρανό αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Ο κοινό ευρωπαϊκό ουρανό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για του λόγου που ήδη αναφέρατε. Ο πιο σημαντικό είναι η συμφόρηση. Μπορούμε λοιπόν να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις όταν δεν επαρκεί ο αναερίος χώρος. Πρέπει να το δούμε έξυπνα. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και με τις προσπάθειες ε, του κυρίου Μαρινέσκου έχουμε μια αρκετά καλή πρόταση. Έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο, αλλά ελπίζω ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί προσεχώς. Αλλιώς δεν θα επαρκεί ο ενέργειος χώρος και έχουμε το εξωτερικό κόστος το οποίο αναφέρατε όπως τις εκπομπές, ε, το χάσιμο χρόνου και μεγαλύτερες αποστάσεις ε, κτλ. Οπότε, με δύο λόγια θα έλεγα ναι, εγώ θα ήθελα να προχωρήσει αυτός ο φάκελος και να το κάνω εγώ και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Σας ευχαριστώ για την απάντηση, κυρία υποψήφια, και μας άρεσε η απάντησή σας, να πω. Γνωρίζετε ότι το μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και ο αντίκτυπος του για το αεροδρόμιο μεταξύ άλλων του Γιβραλτάρ είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ισπανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αεροδρόμιο που έχει οικοδομηθεί σε έδαφος που δεν αναγνωρίζεται ως μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου από τη χώρα μας. Είναι ένα, μία από τις επιπτώσεις που θα έχουμε μέσω του Brexit εφόσον ολοκληρωθεί. Εδώ και χρόνια αναζητούμε μία δίκαιη λύση ώστε να εξυπηρετείται το ίδιο το Γιβραλτάρ αλλά και οι παραμεθόριες περιοχές και πόλεις στην Ισπανία. Νομίζουμε ότι μια λύση θα υποφελούσε και τα δύο μέρη και σας ρωτώ λοιπόν σαφώς κύριε Βαλεάν. Η Επιτροπή θα υπερασπιστεί τα ισπανικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά την αερολιμένα του Γιβραλτάρ. Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε το επίμαχο αυτό ζήτημα. Ελπίζω να βρεθεί στο μέλλον ο καλύτερος τρόπος ε, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Σε αυτή την φάση, στο πλαίσιο του Brexit, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ε, αν συμβεί αυτό, εγώ θα είμαι επίτροπος για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κοφ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαλεάν, έχουμε μια κλιματική ανάγκη. Πρέπει να επιτύχουμε αυτό το 2050 κλιματική ουδετερότητα με ενδιάμεσους στόχους ε, τουλάχιστον 55% μείωση μέχρι το 2030. Παρ' όλα αυτά, οι εκπομπές των μεταφορών αυξάνονται και κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Οπότε, σε σχέση με τα έργα τα οποία δεν ε, είναι θωρακισμένα ως προς αυτήν την πτυχή. Θα τα στηρίξετε. Ο προϋπολογισμός και το προσχέδιο το οποίο υποβλήθηκε λέει ότι υπάρχει μια γενική διάταξη που ισχύει και για τη χρηματοδότηση των μεταφορών έτσι ώστε τα έργα τα οποία δεν συμφωνούν με τους κλιματικούς στόχους δεν θα είναι επιλέξιμα για οικονομική στήριξη και ότι η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις θα ελέγχονται για να οριστεί εάν έχουν κλιματικό αντίκτυπο και αν ναι θα υποστούν την ανάλογη επεξεργασία. Συμφωνείτε λοιπόν να ισχύσουν αυτά για κάθε χρηματοδότηση των μεταφορών της Ένωσης για να επιτυχούμε τον στόχο του 2050 και τους ενδιάμεσους ειδικά δεδομένου του μεγάλου χρονικού ορίζοντα των υποδομών μεταφορών. Ναι, όταν μιλάμε για το κλίμα και τις εκπομπές, όπως βλέπετε αυτό είναι στον πυρήνα των πολιτικών που θα αναπτύξουμε μέχρι το τέλος του επομένου έτους, εάν εκλεγώ, θα παρουσιάσω μια στρατηγική για την βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και το θέμα της χρηματοδότησης των έργων στο πλαίσιο αυτό είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό έγιναν πολλές συζητήσεις για το τι σημαίνει και τι είναι το σωστό που πρέπει να γίνει με οικονομική στήριξη των έργων. και τι χρειάζεται για να ενθαρρύνουμε την ε, έγκριση τέτοιων πράσινων έργων, αν σας κατάλαβα καλά για την μείωση των εκπομπών. Εάν δούμε παραδείγματος χάρη το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, βλέπουμε ότι ένα υψηλό ποσοστό των έργων είναι ήδη πράσινα. 80% νομίζω του φακέλου πηγαίνει σε πράσινα έργα, 72% σε σιδηρόδρομο, 16% σε πλεύσιμους ποταμούς, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Βεβαίως ε, συζητήσαμε την πιθανότητα μιας πράσινης τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη κριτήρια χρηματοδότησης. Νομίζω θα μετασχηματιστεί ε, σε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι επίτροποι θα προσπαθήσουν στο μέλλον να καθορίσουν τα κριτήρια για βιώσιμα έργα αν ήταν αυτή η ερώτησή σας. Ε, είπατε ότι εντάξει, κάπου είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι εκπομπές αυξάνονται σημαντικά και οι ε, μεταφορές είναι εξαίρεση. Και για να αναφερθώ και εγώ στον τομέα της αεροπορίας, γράψατε στις γραπτές σας απαντήσεις πως ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών κατά 10% αλλά θα υπάρξει μια αντιστάθμιση γιατί θα υπάρχει περισσότερο περιθώριο και άρα περισσότερες πτήσεις. Οπότε ίσως υπάρξει σημαντική αύξηση των εκπομπών. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να πετάμε λιγότερο. Συμφωνείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις πτήσεις και όχι να τις αυξήσουμε και να πάμε σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφορών και θα τα πούν αυτά και οι συνάδελφοί μου. Θα δεσμευτείτε στην αρχή ε, ορυπαίνων πληρώνει και για την αεροπορία μέσα μέτρων όπως ο φόρος ο ε, που θέλει ο Φραν Τίμερμανς. Α, είναι Κρίμα που δεν έχω δύο λεπτά στην διάθεσή μου γιατί χρειάζεται πολύ χρόνο. Βεβαίω υπάρχουν όλα τα μέτρα για να απομακρυνθούμε από τι εκπομπέ. Η αποτελεσματικότητα των οχημάτων, τα εναλλακτικά κάψιμα, την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματο. Μετά μιλήσατε για άλλου τρόπου μεταφορών. Οι σιδηρόδρομη Λέω ξεκάθαρα ότι οι σιδηρόδρομη είναι στο επίκεντρο των βιώσιμων μεταφορών και εκεί πρέπει να επενδύσουμε και στη, στα, στις συνδυασμένες μεταφορές. Θέλω τα φορτία να πάνε στα τρένα στο μέτρο του δυνατού. Όταν μιλάμε για την αεροπορία νομίζω η οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται περισσότερες δυνατότητες και ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας, τη μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων Οπότε δεν θα πάω προς την κατεύθυνση του να πω ότι χρειαζόμαστε λιγότερες ε, πτήσεις. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο βιώσιμοι και να έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της εναερίας ε, κυκλοφορίας. Για τον φόρο κυροζήνης ε, θα πω ότι είναι μία από τις πιθανότητες, αλλά πρέπει να είναι σε ένα καλάθι, μια δέσμη μέτρων αγοράς και μη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καμπουμενόζη έχει το λόγο. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Βαλέαν. Εγώ ανησυχώ σχετικά με τις επιπτώσεις κόστους που μπορεί να έχει το Green Deal. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επομένως για τους εργαζομένους. Ιδιαίτερα στην οργάνωση των μεταφορών, όπου έχουμε ήδη σημαντικό μειονέκτημα εναντί μεταφορέων που δεν υπόκειται στις ίδιες διατάξεις στον υπόλοιπο πλανήτη δηλαδή. Έχουμε κοινωνικό dumping εντονότατο από άλλους μεταφορείς και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα συμβαίνει αυτό και μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό σε αντίστοιχε συζητήσει. Σα ρωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρόθεση έχει να κάνει για να υποστηρίξει τι επιχειρήσει των μεταφορών και μιλώ και στις οδικές και στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές και σε συνδυασμό και συνεργασία με τους λιμένες και ιδιαίτερα σε σχέση, επαναλαμβάνω, με το κόστος που θα μπορούσε να είναι πολύ αυξημένο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι ε, απολύτως ουσιαστικό να υποστηρίξουμε την οικονομία διότι ε, στις υπηρεσίες είμαστε από τους παγκόσμιους ηγέτες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προκειμένου να εξαγάγουμε τα δικά μας πρότυπα σε άλλες χώρες. Έχουμε συμφωνίες λοιπόν συνάψη, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις τις δικές μας αλλά και για αυτές που έχουν πρόσβαση στην αγορά μας. Επομένως πρέπει διαρκώς να αξιολογούμε την υλοποίηση των κανόνων αυτών και να δούμε πού βρισκόμαστε. Ε, Μιλώντα για τους λιμένες, θα σας έλεγα ότι η ναυτιλία είναι τεράστιος τομέας, τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι πιο βιώσιμος και πιο πράσινος, αλλά αυτό πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο θετικής ανταπόκρισης, δηλαδή και πιο πράσινος και πιο ανταγωνιστικός. Επί τη βάση ισχυρών διεθνών συμφωνιών, όπου έχουμε τη ρήτρα αυτή της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και των καλών πρακτικών. Με μέτρα και κυρώς προβλέπονται σε περίπτωση καταχρήσεων. Επομένως όλοι οι οικονομικοί φορεί που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας πρέπει να σέβονται τις διατάξεις, του κανόνε που έχουμε εδώ. Και αυτό είναι βασική αρχή της Κομισιόν και θα συνεχίσει να την τηρεί. Ε, κυρία Βάλεαν, ευχαριστώ. Πιο συγκεκριμένα, ένα θέμα που οπωσδήποτε ε, θα σας απασχολεί και θα απασχολεί και τους συναδέλφους σας της εσωτερικής αγοράς ως προς τους λιμένες έχετε αποκλήσεις απόψεων σε σχέση με τις λιμενικές αρχές διότι έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα ε, που θα μπορούσαν να δεχθούν τις, ε, τους ε, λιμενικές αρχές ως ιδιωτικούς φορείς ενώ υπό το Ιταλικό σύστημα είναι ξεκάθαρα δημόσιοι κρατικοί αυτοί οι φορείς. Μπορεί να υπάρξει μια συγχώνευση ή μια, ένα συνδυασμό των δύο αυτών προσεγγίσεων και ένα σύστημα που δεν θα ήταν μειονεκτικό για την Νότια Ευρώπη. Κοιτάξτε, δεν θέλω κανείς να επιβαρυνθεί, κανείς να μείνει πίσω, λέει η κυρία Βάλεαν. Ε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε ενωμένοι, να δουλεύουμε από κοινό και να έχουμε καλή κερδοφορία παντού στην Ευρώπη, λέει η κυρία Βάλεαν. Δεν βλέπω καθόλου ανταγωνισμό μεταξύ περιοχών της Ευρώπης και αν κάπου εντοπιστεί αυτό θα πρέπει να το ε, οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ δεν γνωρίζω τέτοιου είδους ε, αντιπαράθεση αν θέλετε μεταξύ νότιο-ευρωπαϊκών και βόρειο-ευρωπαϊκών λιμένων αλλά στα πλαίσια του μελλοντικού μας ε, συστήματος ναυτιλιακής ανάπτυξης οι λιμένες είναι όχι μόνο κέντρα επιχειρηματικότητας αλλά και έχουν πολύ σημαντικό ίχνος, αποτύπωμα ε, ενεργειακό και επομένως περιβαλλοντικό και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαματίσουν στον, στο πολυτροπικό, πολυ, ε, συνδυαστικό των μεταφορών μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να διατηρηθεί η κερδοφορία τους και πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα με άλλα μέσα μεταφοράς. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Ζήλε, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ και καλώ ορίσατε, κυρία Βαλιάν, στην Επιτροπή Μεταφορών. Καταρχά, θα ήθελα εξ ονόματο του ECR να πω ότι πάντα μπορείτε να υπολογίζετε στι πολιτικέ σα ε, σε ό,τι αφορά στην υποστήριξή μα, αν ε, κινηθείτε προ την κατεύθυνση αυτή που έχουμε επισημάνει. Σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που μα αναφέρατε, έχετε δίκιο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό όμω να μην χάσουμε τα θέματα ουσία για το πώ ε, το Connecting Europe Facility μπορεί να λειτουργήσει σε χώρες ε, της πολιτικής συνοχής κυρίως σε ό,τι αφορά τον ε, τομέα των μεταφορών. Τι σημαίνει αυτό. Θα βρείτε συμβιβασμού μεταξύ του Connect Europe Facility της χώρες του Ταμείου Συνεχής και το πώς θα οργανώσουμε τους τομείς αυτούς. Και μετά από αυτά που ακούσαμε εδώ θα υπάρχουν λιγότερες πτήσεις, αλλά Υπάρχουν ακόμα χώρες που δεν συνδέονται σειροδρομικά με άλλες χώρες. Όλες αυτές τις ψηλολεπτομέρειες θα τις ε, υποστηρίξετε προκειμένου να ρυθμιστούν πρώτου μάλιστα ολοκληρωθεί και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση του δικτύου TNT είναι απολύτως απαραίτητη. Προφανώς ε, έχει καθυστερήσει, αλλά Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπιση ε, του θέματο. Το 2021 επίση θα αναθεωρήσουμε και τι κατευθυντήριε γραμμέ για τα δίκτυα TNT. Ξέρω ότι υπάρχει τη σχετική δέσμευση. Θα δούμε λοιπόν τι χρειάζεται για να υπάρξει σχετική αναβάθμιση. Κοιτώντα το χάρτη τη Ευρώπη, βλέπουμε τεράστιε διαφορέ στην ε, συνδεσιμότητα, στην διασύνδεση μεταξύ Ανατολή και Δύση. Ξέρω ότι αν κανείς τα έχει όλα μπορεί να πει ότι κοιτάξτε με την εμπειρία μας μπορούμε να αποφύγουμε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι παρόλα αυτά η Ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να τύχει πλήρω υποστηρίξει για να αναπτύξει ένα συνεκτικό και πλήρε δίκτυο και θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευφύοι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο Connecting Euro Facility, ήθελα να τονίσω και να προωθήσω τις συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων τομέων. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν ένα ευφύ χαρακτήρα προκειμένου να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε διάφορα εργαλεία να αναπτυχθούν εκ παραλλήλου. Λύσεις μεταφορών, ε, ψηφιακές λύσεις για παράδειγμα, συνεργασίες και συνέργειες με άλλους τομείς για την ε, ολοκλήρωση του δικτύου, του κεντρικού δικτύου, προάσπιση των πόρων ε, συνοχής και να έχουμε υπόψη ότι η σιδηρόδρομη είναι η πιο καθαρή μόρφη μεταφοράς, άρα με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να συμβάλλουμε σε όλα τα έργα στον κλάδο αυτό. Η Επιτροπή αυτή, στην Επιτροπή αυτή ξέρετε ότι εργαζόμαστε για το πακέτο κινητικότητας 1 και 2. Για το πρώτο πακέτο κινητικότητας ξέρετε ότι έχουμε έξι πρωθυπουργούς που έγραψαν μια επιστολή στην Επιτροπή με τις ιδέες αυτές και ότι έχουν χάσει τον αρχικό τους στόχο. Ίσως να πετύχουμε μια συμφωνία πριν να λάβετε καθήκοντά σας. Θα δούμε λοιπόν όμως ε, τα αποτελέσματα. Είσαστε διτεθειμένοι να κάνετε μια μελέτη αντικτύπου και αν προκύψει κάτι θα χρειαστεί να το διορθώσουμε να το κάνουμε για το δεύτερο πακέτο κινητικότητα τώρα. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοβουλία της κυρίας Μπούλτσα. Θα προωθήσετε λοιπόν τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο για να κινηθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητα 1 και 2 στο Συμβούλιο. Η απάντηση. Κοιτάξτε, για το πακέτο κινητικότητα πιστεύω ότι είναι απολύτω απαραίτητο να εγκριθεί για να μην ξεχνάμε γιατί προτάθηκε. Γιατί χρειάζεται και η εσωτερική αγορά να λειτουργεί καλά. Και καλές υπηρεσίες για τους εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εγκριθεί, είναι ύψη τη σημασία. Ελπίζω να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζω και πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Από την άλλη, να πω το εξή. Σε κάθε νέα νομοθεσία που προκαλεί διχασμό, θα κληθούμε να κάνουμε αξιολόγηση και να συζητήσουμε μαζί σας κατά πόσον υπάρχει περιθώριο βελτίωσης μέσω επιπρόσθετων μέτρων. Αυτό σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η σχετική διάταξη, γιατί αν αυξηθεί ο αριθμός λεωφορείων και πούλμαν, αυτό θα έχει σαφή πλέον εκτίματα. Γιατί έτσι θα μειωθούν οι επιβάτες σε άλλα χερσαία οχήματα και θα μειωθεί και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοντουρά έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την υποψήφια Επίτροπο για την πλήρη εισαγωγική της τοποθέτηση. Η εντολή που έχετε λάβει από την Πρόεδρο της Επιτροπής είναι πραγματικά πολύ φιλόδοξη και επικεντρώνεται στο μετασχηματισμό του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο του European Deal, Green Deal και με στόχο τη μηδενική ρήπανση. Μα είπατε ότι και εσεί συμμερίζεστε αυτό το στόχο και μα αναφέρατε τι προτεραιότητέ σα. Θα θέλαμε να μάθουμε λοιπόν ε, πώ θα τι υλοποιήσετε. Θέλω να σταθώ σε μια πολύ σημαντική διάσταση του μετασχηματισμού του συστήματος μεταφορών που πολύ συχνά ξεχνάμε. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο μετασχηματισμό θα γίνει χωρί αποκλεισμού κυρίω των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και των πιο απομονωμένων νησιωτικών περιοχών, διότι ξέρουμε ότι ο μετασχηματισμό θα έχει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα ένα τεράστιο κόστο, το οποίο δεν είναι ακόμα σαφέ πώ θα κατανεμηθεί. Οι οικονομικά ισχυροί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, ενώ στι νησιωτικέ περιοχέ το κόστος των μεταφορών επιβαρύνει ήδη δυσανάλογα τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι πιο ευάλωτοι στις κοινωνίες μας θα έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές μεταφορές άμεσα αλλά και έμεσα στην περίπτωση των εμπορευμάτων. Αυτά τα δύο θα πρέπει να πάνε Γιατί χρειαζόμαστε και πολυτροπικέ μεταφορές και νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και χρόνο και χρήματα και προσπάθεια για να τα πετύχουμε αυτά. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αυτό θα είναι προ όφελο των μεταφορών, των επιχειρήσεων, προκειμένου να μετακινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή οι επιχειρήσεις μας, να μπορέσουν να μετακινούνται με πιο γρήγορο τρόπο και με πιο χαμηλό κόστος. Το γεγονός ότι υπάρχουν απομονωμένες περιοχές και ότι εκεί χρειάζεται ειδική μεταφορά. Ξέρω φυσικά ότι ζεστεύετε την Ελλάδα και το θέμα αυτό το κατέχετε ιδιαίτερο γιατί η Ελλάδα έχει τεράστιο αριθμό νησιών. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν ζήτημα. Σημαντικό πρόβλημα. Η διασύνδεση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να επενδύσουμε για να είναι συνδεδεμένες αυτές οι περιοχές με βιώσιμο τρόπο γιατί ξέρουμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδος που είναι τουριστικός προορισμός ε, και ο τουρισμός θα πρέπει να έχει ένα δίκτυο υποδομών. Το θέμα λοιπόν της διασύνδεσης παραμένει το πιο σημαντικό στοιχείο. Θα επενδύσουμε στη διασύνδεση. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα αεροδρόμια και τα τοπικά αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζονται όλα αυτά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε. Εκτός μικροφώνου. Ναι, ακούγομαι. Σχετικά με τη ρήπανση που προέρχεται από την αυτιλία και ειδικότερα στα λιμάνια, πιστεύετε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για τη χρήση υγροποιημένου αερίου και για μια ε, και από ξηρά παροχή ηλεκτρική ενέργεια. σκοπεύετε να αξιολογήσετε τη σκοπιμότητα μια λύση, όπω παραδείγματο χάρη στην Καλιφόρνια που υπάρχει υποχρέωση για τα πλοία και πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εγκαταστάσει για αποξηράς ηλεκτρική ενέργεια και συγκεκριμένου φιλόδοξου στόχου για τη χρήση αυτή τη τεχνολογία. η εχετε καποιο αλλο σχεδιο όπω για παραδειγμα η προωθηση του υδρογόνου εναλλακτικά. Και ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα για την επιστολή που έστειλε η πρόεδρός μας, η κυρία Ντέλη, στην ε, πρόεδρο, την κυρία Βόντε Λάιεν, με την οποία ζητούσε τη δημιουργία χαρτοφυλακίου στη Νέα Επιτροπή, όπου οι μεταφορές θα είναι μαζί με τον τουρισμό. Όπως γνωρίζετε, η σημασία του τουρισμού είναι τεράστια, είναι το 10% του ΑΕΠ της Ευρώπης, το 11% των θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από αυτόν και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς μεταφορές και μεταφορές χωρίς τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you for the question. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Το θέμα της θαλάσσιας ρήπανσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρουμε ότι τίθεται και το θέμα της ρήπανσης της ατμόσφαιρας λόγω ε, των ε, οξυδίων αζότου. Και ξέρουμε επίση ότι τα απορρίμματα, τα θαλάσσια, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για τον πλανήτη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και σχετική οδηγία, την οποία θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να αναπτυχθούν σχετικέ εισαγωγέ και υποδομέ για εισαγωγέ εναρκτικών καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή του coming plug-in για την η ηλεκτρική ενέργεια για τα πλοία στα λιμάνια. Υπάρχει επίσης και μία ιδέα για τα πράσινα πλοία. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω για να γίνει πιο πράσινη και η ναυτιλία. Για τα λιμάνια και για την θαλάσσια ρηπανσή. Ένα από τα εργαλεία που υπάρχουν Μία από τις ευκαιρίες είναι και η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Βιοπικιλία, προκειμένου να εστιαστούμε πιο πολύ στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Υπάρχουν λοιπόν νομοθετικές, νομοθετικά εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε πώς εφαρμόζονται, πώς υλοποιούνται και πώς μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Euh, Ευχαριστώ τελευταία ερώτηση σε αυτόν τον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Το λόγο έχει. Έχουν ε, ολοκληρώθηκε μάλλον η πρώτη, ο πρώτος γύρος και τώρα θα πάρουν το λόγο οι βουλευτές για το δεύτερο γύρο. Το λόγο έχει η κυρία τελεία; Ένα λεπτό. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βαλεάν, αναφέρατε το σιδηρόδρομο πριν από λίγο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο κλάδος ε, πρέπει να, επιτύχει το πλήρες δυναμικό του. Ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ βασικός για να συμβεί αυτό, να γλιτώσουμε εκπομπές και χρήμα. Ποιες προτάσεις συγκεκριμένα θα κάνετε ως Επίτροπος για να ανοίξει η αγορά του σιδηρόδρομου, για να έχουμε υγιή ανταγωνισμό και ποιοτικέ υπηρεσίες και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της διαλειτουργικότητας και πώς θα διασφαλίσετε την ε, χρηματοδότηση ε, της εφαρμογής του ERTMS, ε, του συστήματος σήμανσης. Ευχαριστώ κυρία Τάλερ. Πρέπει να εφαρμοστεί το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Είναι πολύ σημαντική η σιδηροδρομή για τις βιώσιμες μεταφορές, αλλά πρέπει να βελτιωθούν δραστικά, γιατί θα πρέπει βεβαίως να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή σιδηροδρομική περιοχή. Να έχουμε νέες τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα για τα δρομολόγια και οπωσδήποτε το νέο σύστημα σήμανσης. Μόνο έτσι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες ε, και αξιοπιστία του συστήματος. Όπως είπα έχουμε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο με τους δύο πυλώνες, τον πυλώνα της αγοράς και τον τεχνικό πυλώνα και χρειάζεται εφαρμογή αφενός μέσω του πυλώνα της αγοράς θα πρέπει να βελτιώσουμε παραδείγματο χάρη την πρόσβαση στις ε, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και εδώ πέρα χρειάζεται. Παραδείγματο χάρη ο εξυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων για να γνωρίζουμε ποιε είναι οι δυνατότητε αυτών των εγκαταστάσεων. Να δούμε το θέμα του τροχαίου υλικού, των εισιτηρίων, για να μην υπάρχουν προβλήματα στην διανομή. Από την άλλη, εάν δούμε τους διαδρόμους ε, και τον σχετικό κανονισμό για το σιδηροδρομικό φορτίο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε προσεκτικά την εφαρμογή και να δούμε τους φραγμούς που υπάρχουν ακόμα στην αγορά από τον κατακαιρματισμό εθνικών κανόνων, από την, ε, τα διασυνοριακά τέτοια εμπόδια, το διεθνές εμπόριο αγαθών, ε, τα οποία όταν διασχίζουν τα σύνορα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες Όλα αυτά υπάρχουν στο τέταρτο πακέτο, πρέπει να εφαρμοστεί. Και θα πρέπει ακριβώ. Ε, ε, παρακαλώ, ολοκληρώστε, λέει ο πρόεδρο. Να δούμε πώ μπορεί να βελτιωθεί ο κανονισμό. Σα ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτησή μου αφορά την επιβολή. Πώς θα επιβάλλετε την συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και θα ξεκινήσετε διαδικασίε επί παραβάση κατά κρατών μελών εάν αυτό απαιτείται. Νομίζω η απάντηση είναι προφανής ε, και περιέχεται στην ερώτηση. Ε, Βεβαίω ε, δεν έχει νόημα να γράφουμε νόμους χωρίς να τους εφαρμόζουμε. Ξέρω βεβαίως πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά εκεί όπου δεν προχωράνε τα πράγματα Οπωσδήποτε θα φέρουμε διαδικασίες επί παραβάση. Παραδείγματος χάρη για τον τεχνικό πυλώνα έχουμε ε, ορθές πρακτικές γιατί έχουμε 8 κράτη-μέλη πρέπει να έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο μέχρι το 2019, μέχρι τον Νοέμβριο. Οπότε το κοιτάμε αυτό. Αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη επέλεξαν να μεταφέρουν τον ε, τεχνικό πυλώνα ε, μέχρι τον Ιούνιο του 20. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι άλλος ένας έτος ε, βεβαίως θα δώσει τη δυνατότητα στην νομοθεσία να οριμάσει. Σας ευχαριστώ. Και το λόγο το έχει ο κ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρία Βαλιάν. Η Ursula von υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, πρότεινε νομοθεσία για να αυξηθούν ε, οι στόχοι μείωση των εκπομπών κατά 50% κατά 55% αν είναι δυνατόν. Και πριν από τρει εβδομάδε, ε, το πολιτικό σα ανέφερε, σα παρέθεσε ότι είπατε το εξή. Δεν θέλουμε να υπάρξουν αλλαγέ σε αυτή την νομοθεσία σε ό,τι αφορά τους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα μέχρι το 2030. Είσαστε λοιπόν ε, δεσμευμένοι στους στόχους που προτείνει η κυρία Φοντερ Λάιεν ή αυτά που λέει η νομοθεσία. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά. Απάντηση. Αυτό είναι λίγο εκτός ε, του συγκεκριμένου πλαισίου. Αλλά να απαντήσω το, εξή. το εξής. Σας είδα και στους τριμερείς διαλόγους ε, να αγωνίζεστε για ένα συνεκτικό και ευρύ πακέτο για την περιορισμό των εκπομπών. Έχουμε δει λοιπόν πόσο σημαντικό και πόσο δύσκολο ήταν να καταφέρουμε μια συμφωνία για τους κανόνες. Το πακέτο για την καθαρή ενέργεια εγκριθήκε φέτος και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής δεν είναι καλό για τις επιχειρήσεις και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που χρειάζονται για τις υποδομές να αλλάζουν οι στόχοι λιγότερο από ένα έτος πριν την εφαρμογή τους. Μετά την εγκρισή τους. Αυτό είναι το πρώτο το μήνυμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια προβλεψιμότητα σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Από την άλλη, προφανώς και πρέπει να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε. Αυτή είναι η αποστολή που μου εμπιστεύεστε μαζί με τον ε, Επίτροπο Τίμερμαντς και τους άλλους επιτρόπους για να βρούμε ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να προσθέσουμε και άλλα επίπεδα σε ό,τι αφορά την ε, περιορισμό των εκπομπών με την εφαρμογή νομοθεσιών σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του συστήματος εμπορίας ρήπων στις θαλάσσιες μεταφορές Πολλά μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του συστήματος επισήμανσης. Αυτό θα δημιουργήσει ένα σύστημα μεταφορών πιο αποτελεσματικό, με πιο καλά κίνητρα για πολυτροπικότητα και αυτή την αλλαγή θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ευθύς αλλαγή. Έχουμε τις κοινοπραξίες, έχουμε την αποτελεσματικότητα των οχημάτων, έχουμε την ανάπτυξη του στόλου των οχημάτων. Έχουμε εναλλακτικέ μορφέ κινητικότητα και υποδομέ σχετικέ. Να αλλάξουμε επίσης και την συμπεριφορά των καταναλωτών για πιο καθαρές λύσεις και στις μεταφορές. Έχουμε λοιπόν ένα καλάθι εργαλείων. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι το οποίο κρίθηκε πριν από κάποιους μήνες. Αυτό το μήνυμα ήθελα να μεταβιβάσω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για τον κατάλογο αυτών των ενδεχόμενων και πιθανών μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν αμφισβητείτε του συνολικού στόχου που προτείνει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Δεν του αμφισβητώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πολύ σύντομα τα καταφέρατε. Ναι, ναι συνεννοούμαστε καλά, λέει η κυρία Βαλεάν. Λοιπόν, η κυρία Νάκτεγκαλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σύστημα ITS για τον τομέα των θαλασσομεταφορών, μεταφορών, η ε, Κομισιόν, η Επιτροπή της κυρίας Φοντερ Λάιεν θέλει να σε πιο βιώσιμο τον κλάδο αυτό. Όλα αυτά είναι σαφή και ευλόγα. Κοιτώντα ε, τον κλάδο αυτό, βλέπουμε ότι δεν τα λένε μόνο αυτά τα πράγματα, αλλά τα κάνουν και όλα τα υλοποιούν. Και είναι πολύ σημαντικό να συμβούν όλα αυτά. Ο ναυτιλιακός ε, κλάδος ε, άλλωστε είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αν υπάρξουν ε, νομοθεσία πιο αυστηρή, θεωρώ ότι θα είναι σε μηνεκτική θέση ο ευρωπαϊκός κλάδος. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι η επίτροπο αυτά θέλει να επιδιώξει. Ερωτώ μήπω θα ήταν ε, πιο λογικό η βιωσιμότητα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών να γίνει μέσω του Διεθνούς ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού προκειμένου ο δικός μας ο κλάδος να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ναυτιλιακό κλάδο, ο, ε, ο κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια μείωση των εκπομπών. Για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε και να διατηρήσουμε και την ηγεσία μας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και την αξιοπιστία μα σε τελική ανάλυση. Φυσικά, οι θαλάσσιε μεταφορέ αποτελούν παγκόσμιο ζήτημα και εμεί λειτουργούμε σε αυτό το παγκόσμιο συγκείμενο έγιναν προσπάθειες, ξέρω, να προωθηθεί αυτό το όραμα που υπάρχει σε επίπεδο διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Και χαίρομαι που για πρώτη φορά ακούσαμε και ένα αριθμητικό στοιχείο στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Μείωση 50% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 με μεταρρύθμιση και αναθεώρηση το 2023 σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε σε επίπεδο IMO για να υπάρξει μία έγκριση σαφών μέσων σε ό,τι αφορά και το δικό μας όραμα θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στα πλαίσια του IMO. Διαρκώς λοιπόν μετακινούμαστε, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Εμείς θα πρέπει να τους πείσουμε να κάνουν αυτό το βήμα πιο γρήγορα. Η Ευρώπη μόνο μερός μπορεί να έχει ειδικά της ε, μέτρα. Θα είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά θα επιδείξει ηγεσία εδώ η Ευρώπη. και το σύστημα εμπορία ρήπων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θεωρώ ότι είναι απολύτω απαραίτητο. Γιατί και οι θαλάσσιες μεταφορές εξαιρούνταν ως τώρα ενώ όλοι οι κλάδοι συνέβαλαν. Και προφανώς είναι και παγκόσμιος αυτός ο κλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία προσωπική ερώτηση. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι το σύστημα ETS εμπορίας ρήπων δεν θα αποβεί εις βάρος των ίσων όρων ανταγωνισμού ε, στον τομέα των μεταφορών και δεν θα υπάρξει ε, θέμα διαρροής άνθρακα από μη ευρωπαϊκές χώρες και αν μπορείτε να μας υποσχεθείτε πώς θα το πετύχετε. Καταρχάς, το πρώτο βήμα είναι να γνωρίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όταν θα αναπτύξουμε το σύστημα εμπορίας ρήπων για τις θαλάσσιες μεταφορές, αν και προφανώς έχουμε προφανώς ε, πολλή εμπειρία από τους άλλους τομείς στους οποίους ε, εργαζόμαστε και προφανώς και διαρροή άνθρακα αποτελεί ε, σημαντικό θέμα. Όταν όμως θα υποβάλουμε την νομοθετική αυτή πρόταση, θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστικότητα του κλάδου, γιατί αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστοφ Χάνσεν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί κυρία Βάλεαν, στις αερομεταφορές έχουμε 25 και άνω αύξηση των εκπομπών στα τελευταία, στην τελευταία δεκαετία. Επομένως πρέπει να επιτυχθούν πρωτοβουλίες ώστε οι αερομεταφορές στην Ευρώπη να γίνουν πιο καθαρές. Ως οριστής επίτροπος λοιπόν πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα δοθούν κίνητρα για τα συνθετικά καύσιμα μεταξύ άλλων που θα πρέπει να φτάσουν μέχρι και τους αερομεταφορείς και να χρησιμοποιηθούν. Κοιτάξτε, όταν μιλώ για πιο βιώσιμο και πιο καθαρό κλάδο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλη τη δέσμη μέτρων της αγοράς και εκτός αυτών. Θα πρέπει δηλαδή να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αντιστάθμισης κλιματικής ε, τη κλιματική αλλαγή, τη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της υποστήριξη της οικονομίας και τη ανταγωνιστικότητας όπως και των χαμηλών τιμών. Από το καλάθι αυτό μέτρων, λέει η κυρία Βάλεαν, έχουμε το ETS, έχουμε το Corsia, για να μειώσουμε τις εκπομπές, θα έχουμε το Κόρσια που όταν θα υιοθετηθεί θα πάμε να το υλοποιήσουμε ώστε να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στο σχεδιασμό των αεροσκαφών και την τεχνολογία τους για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στα αεροκαύσιμα, καλύτερη διαχείριση της ε, εναέριας κυκλοφορίας, ε, εξοικονόμηση καυσίπου και βιώσιμα καύσιμα που αναφέρατε κι εσείς. Αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά κόστους τιμής μεταξύ κυροζίνης και άλλων καυσίμων. Κάτι που φαίνεται να είναι ελπιδοφόρο, είναι η χρησιμοποίηση προς το παρόν μειγμάτων ε, καυσίμων, αεροκαυσίμων. Θα πρέπει μακροπρόθεσμα να έχουμε βιώσιμα καύσιμα, δεν είμαστε ακόμα εκεί αλλά έχουμε κάποια έργα που φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές για το μέλλον και στην μετατροπή από βιώσιμες ε, πηγές ενέργειας, ηλιακή προς καύσιμα για παράδειγμα, είναι νέες τεχνολογίες που πρέπει να διερευνήσουμε, ε, να ερευνήσουμε περαιτέρω για να δούμε πού μπορούμε να οδηγηθούμε και τι μπορούμε να πετύχουμε ώστε να είμαστε και φιλικοί προς το περιβάλλον, αλλά να μην απολύσουμε και ανταγωνιστικότητα. Ναι, να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα μεταξύ διαφόρων καυσίμων. Ποιες είναι οι σκέψεις σας ε, για την οδηγία, για την φορολόγηση των καυσίμων. Ε, βέβαια γνωρίζουμε ότι μπλοκάρουν αρκετά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και γι' αυτό δεν προχωρεί, αλλά βλέπετε κανένα περιθώριο μόχλευσης τέτοιων ειδικών φόρων επί των καυσίμων και θα μπορούσε ένας νέος ευρωπαϊκός φόρος να κατευθυνθεί απευθείας στους, στους ίδιους πόρους ώστε ακριβώς να αντισταθμίσει την κλιματική αλλαγή. Ε, ναι, ακριβώς ε, το πρόβλημα είναι πού πηγαίνουν τα φορολογικά είσοδα. όπως λέτε κι εσείς, γιατί μετακυλίονται και στο, στην τιμή του εισιτηρίου και στους καταναλωτές. Πόσο αποτελεσματικός λοιπόν θα ήταν ένας τέτοιος φόρος οικονομικά και κοινωνικά. Θα, θα έπρεπε κανείς να ερευνήσει. Γνωρίζω ότι κάποια κρατημέλη ήδη εφαρμόζουν τέτοια επιβάρυνση Μάλιστα λέγεται ότι εξετάζεται και η νομοθεσία του ΦΠΑ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά και να σκεπτόμαστε πάντα το σύνολο του καλάθου των μέτρων. Και να λάβουμε υπόψη μας και άλλες τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκαρθία Μουνιώθ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, γνωρίζετε οι μεταφορές ε, είναι πολύ μακριά από το να έχουν επιτύχει η ισότητα των φύλων. Έχουμε ιδιαίτερα έντονη εκπροσώπηση των ανδρών και αναφέρομαι στο θέμα της ισότητας των φύλων στην εργασία. Η πλατφόρμα γυναίκες στις μεταφορές θα επηρεάσει την μελλοντική στρατηγική της Επιτροπής αλλά κυρίως μπορείτε να μου πείτε τι νομοθετικά μέτρα συγκεκριμένα και απτά έχετε την πρόθεση να αναλάβετε ώστε να εξασφαλίσετε υψηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των μεταφορών για να έχουμε ίσες ευκαιρίες όπως και μισθολογικές αποζημιώσεις. Επίσης, ποια μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε για την επανακατάρτιση του γυναικείου ε, προσωπικού, ιδιαίτερα εκείνου της μέσης ηλικίας. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ήδη σχολίασα ότι ήθελα να εργαστώ προς ένα τομέα πιο ισόρροπο μεταξύ των φίλων. Γνωρίζουμε το ο τομέας αυτός κυριαρχείται από τους άνδρες, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε λήψεις στο προσωπικό. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να το καλύψουμε, βλέποντας και τι εργαζόμενους θέλουμε να προσελκύσουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν το τομέας να είναι ελκυστικός και για νεότερους ανθρώπους και για γυναίκες και για πολλεπλών εθνικοτήτων ανθρώπους, δηλαδή για να προαγάγουμε τη διαφορετικότητα, πιστεύω ότι Εάν τα καταφέρουμε θα έχουμε πιο ανταγωνιστικό συνολικά τομέα λόγω ακριβώς της συνεισφοράς της διαφορετικότητας των ανθρώπων που θα εργάζονται εκεί. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη γύρανση του συνολικού προσωπικού. Όπως επίσης πρέπει να δουλέψουμε για την εικόνα, το image του τομέα και επομένως και τις συνθήκες εργασίας. ώστε να προσελκύουμε νέους εργαζομένους στον τομέα. Ε, γνωρίζω ότι ο Επίτροπος Μπούλς είχε δουλέψει επί της πλατφόρμας αυτής για τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επέλθουν στον τομέα και είναι ένας τρόπος για να καταστήσουμε τον τομέα πιο ελκυστικό που σας έλεγα και να αλλάξουμε το θεματολόγιο. Έχουμε και την Επίτροπο Ντέλη για τα θέματα ισότητα των φύλων και άλλου συναρμόδιους που θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα στο δικό τους πεδίο, αλλά ε, είμαι βέβαιη ότι θα αναλάβουμε πολλές δραστηριότητε σε επίπεδο συνολικά της Επιτροπής, ώστε να υποστηρίξουμε την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών και εσωτερικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο λέει η κυρία Φάλεα. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και μιλώντας για ίσες ευκαιρίες και βελτίωση των συνδικών εργασίας, όπως και εσείς λέγατε, ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, οι συνθήκες απασχόλησης και οι συνθήκες ασφάλειας στις αερομεταφορές ιδιαίτερα ε, απαιτούν νομοθετικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων στον τομέα και η ασφάλειά τους. Και γι' αυτό σας ρωτώ τι μέτρα πρόκειται η Επιτροπή σε συνδυασμό με την ε, μαζί με την ΕΑΣΑ ώστε να εξασφαλιστούν δίκαιες συνθήκες εργασίας κοινωνικέ συνθήκες για του ανθρώπου συνολικά που θα εργάζονται στον τομέα αυτό και τους επιβάτε. Ε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιη, λέει η κυρία Βάλεν, ότι αντελήφθη απολύτως καλά την ερώτησή σας. Εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες εργασίας είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό σε οποιονδήποτε τομέα. Και βεβαίως η ασφάλεια επηρεάζει άμεσα το αίσθημα της ασφάλειας. Επηρεάζει άμεσα το πώς εργάζονται καθημερινά οι άνθρωποι στον τομέα. Υπάρχουν ανάγκες οικογενειακές που θα πρέπει να καλύπτονται προκειμένου να ε, ε, παραμένει ελκυστικός ο τομέας και να έχουμε μια καλύτερη σύνθεση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στη διάθεσή μα δηλαδή καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αλλά και πάλι λέω δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα τι ρωτούσατε. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ντεπαρνέ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλεάν, εδώ και 150 χρόνια η σιδηροδρομή είναι το μεταφορικό μέσο το πιο φιλικό προς το περιβάλλον και τους χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Γι' αυτό αναρωτιέμαι για την απουσία του σιδηροδρόμου από την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων αλλά και από την ομιλία σας σήμερα. Δυστυχώς η πολιτική μεταφορών αδικοί τους ε, σιδηροδρόμους. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, παραδείγματος χάρη η αρχή όροι πένων πληρώνει. Δεν εφαρμόζεται παρκώς για τις οδικές μεταφορές. Ο ΦΠΑ ισχύει για τις ε, διασυνοριακές, τα διασυνοριακά δρομολόγια σιδηροδρόμου, αλλά όχι για τις πτήσεις. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφορά και να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη θα επενδύουν περισσότερο σε σιδηροδρομικές υποδομές. Αυτές είναι βασικές απαιτήσει για να αλλάξουμε μέσα μεταφορά, Υπάρχει ο σιδηρόδρομος στην επιστολή εκεί που λέει ε, μια στρατηγική για βιώσιμες ε, μεταφορές. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να ευνοήσουμε τις επενδύσεις τους ε, σιδηροδρόμους και να επενδύσουμε στην διατροπικότητα για να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους. Θα έλεγα πως ε, υπάρχουν αυτά εκεί μέσα. Τώρα. Τι άλλο με ρωτήσατε. μέλλον. Ανταγωνιστική σιδηρόδρομη, ναι. Όπως είπα έχουμε το πακέτο το σιδηροδρομικό, έναν καλό πυλώνα αγοράς και έναν τεχνικό πυλώνα. Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε τον κατακαιρματισμό, τους διάφορους εθνικούς κανόνες. Αλλά δεν ξέρω, μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας γιατί δεν το συγκράτησα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ο οικολογικός μετασχηματισμός σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές. Αν θέλετε να δείτε τις εκπομπές των φορτηγών, πρέπει οι μεταφορές να πάνε στα τρένα. Ε, και για τα αεροπλάνα επίσης πρέπει να ξαναφέρουμε τα νυχτερινά τρένα για να υπάρχουν εναλλακτικέ. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμώ αυτό το οποίο είπατε ότι η αγορά των εισιτηρίων των τρένων και η αλλαγή εταιριών πρέπει να γίνει πιο εύκολα αλλά ο σιδηροδρομός θα αναπτυχθεί πλήρως όταν υπάρχει δικτύωση και επιλογές. Οπότε θα κάνω τώρα την ερώτησή μου. Ποια είναι τα σχέδιά σας για να διασφαλίσετε την συμπερίληψη διασυνοριακών νυχτερινών τρένων. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, με είχατε ρωτήσει πριν για το εξωτερικό κόστος των οδικών μεταφορών και προτεραιότητα θα ήταν να ενσωματωθεί αυτό το κόστος, οπότε ε, υπ' αυτό το πρίσμα συμφωνώ μαζί σας, βεβαίως προσεκτικά, γιατί η εξωτερικεύση του κόστους δεν είναι το μόνο μέσο που έχουμε και μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες άλλες συνέπειες. Για τα φορτία μέσω στυροδρομού πρέπει να πάνε τα εμπορεύματα με το τρένο, απλό είναι. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στις υποδομές, στην διατροπικότητα, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα εμπόδια Και παραδείγματο χάρη ναι, ε, κάτι το οποίο μας εμποδίζει σε τέτοια τέρμιναλ ε, είναι διάφοροι φραγμοί που υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ψηφιοποίηση έτσι ώστε τα αγαθά όταν αλλάζουν μέσω μεταφοράς ε, να είναι τα πάντα ψηφιοποιημένα τα έγγραφα. Τώρα είναι όλα χάρτινα και αυτό είναι απαράδεκτο. Εξυγχρονισμός λοιπόν, καινοτομία πολλαπλά μέσα μεταφοράς ε, για να πάνε τα φορτία στα τρένα. Και κάτι άλλο, εγώ είμαι υπέρ των νυχτερινών τρένων, αρκεί να είναι ανταγωνιστικά. Και βεβαίως ε, εκεί πέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλίπ Ολιβιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλεάνα. Λέτε ότι θα πρέπει να ε, πετύχουμε ένα στόχο ε, ανθρώπινο και οικολογικό. Δεν έχουμε ακόμα μιλήσει για τους εργοδότες. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο το οποίο θα προωθήσει με τέτοιο τρόπο τις ε, μεταφορές. Πιστεύετε ότι μπορούμε να πετύχουμε με βιώσιμο τρόπο τέτοιες ηλιακές μορφές ενέργεια, για παράδειγμα. Μπορούμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, μπορούμε να γνωρίσουμε τις ανθρώπινες κοινότητες. Ως ε, Ρουμάνα, πώς θέλετε να αντιμετώπισετε το θέμα των αποσπασμένων εργαζόμενων, που ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχετε ιδιαίτερα στην πατρίδα σας, ε, που ζουν μακριά από τον χώρο που δουλεύουν. Και πώς μπορείτε να πετύχετε η κυβέρνησή σας να αντιμετωπίσει θέματα όπω για παράδειγμα οι Πακιστανοί που εργάζονται κατά χιλιάδε ή δεκάδε χιλιάδε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα οικολογικά και ανθρωπιστικά τα οποία θέτονται και πολλά μερικατελεστικά στοιχεία τα οποία διακρίνονται στην πολιτική σα. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι και Ρουμάνα και ε, υπέρ του ουμανισμού, του ανθρωπισμού. Δεν βλέπω την αντίθεση. Και όπως είπα στην αρχή, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία του, της βιώσιμης κινητικότητας. Όταν μιλάτε για τις συνθήκες εργασίας, για το πακέτο κινητικότητας προφανώς, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο νομοθετικό πακέτο, κάποιο άλλο νομοθετικό πλαίσιο. που να διχάζει το Κοινοβούλιο τόσο πολύ όσο το πακέτο γεννητικότητα. Γιατί προφανώ αφορούσε υπερβολικά πολύ κάποιε χώρε, κάποιε ιστορικέ αγορέ, κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάποιου. Ενώ θα έπρεπε να έχει εστιαστεί στην καλά καλή ενιαία αγορά και στις καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αυτό υποστηρίζω. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλό αποτέλεσμα του πακέτου κινητικότητας προκειμένου να έχουμε και τις δύο πτυχές. όπως και οι συνάδελφοι και εγώ έχω να παρατηρήσω ότι δεν είσαστε πολύ συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά μέτρα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτό να μην αποτελεί προτεραιότητά σας. Μια ερώτηση λοιπόν να σας κάνω ακόμα. Θα παρέμβετε σε ό,τι αφορά τους αποσπασμένους, ε, σε ό,τι αφορά τα... την επιβάρυνση που δέχονται. Και τις ε, απάτες. Είπατε απάτες κατάχρηση σε ποιο σκέλος. Φυσικά θα ήθελα να καταπολεμήσω την ε, απάτη και τις καταχρήσεις. Ε, ποιος δεν θα ήθελε αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Θέλω να συνεργαστώ με του ε, συναδέλφου μου, τους άλλους επιτρόπους, για να αναλάβουμε δράση σε όλους αυτούς του τομεί προκειμένου οι εργαζόμενοι. Και το εργασιακό περιβάλλον στον τομέα του, των μεταφορών να προστατευτεί από τις απάτες, από τις καταχρήσεις. Αυτή είναι η στάση μου. Σας διαβεβαιώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την δήλωση που κάνατε ότι ε, θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Αναφέρατε πόσο διχαστικό ήταν ε, στην προηγούμενη θητεία το πακέτο κινητικότητας. Η ερώτησή μου τώρα, τι θεωρείτε ήταν το πιο επικίνδυνο κομμάτι αυτού του πακέτου. Η επόμενη μου ερώτηση αφορά επίσης ε, την αεροπορία, τον μόνο κλάδο που δεν ε, περιλαμβάνεται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Τώρα όμως έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα και φαίνεται ότι και τα δύο συστήματα αυτά θα λειτουργήσουν παράλληλα. Θα καλύπτεται λοιπόν η αεροπορία από τα συστήματα αυτά. Και βεβαίως μιλήσαμε για τα διευρωπαϊκά δικτύα, για την κινητικότητα, για το ποια, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο για εσάς, για την επιτροπή σας, όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του συστήματος αυτού. Ναι, ε, δεν θέλω να αναφερθώ στο πακέτο κινητικότητας, γιατί για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη φάση είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου. Είναι σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να αναφέρω εγώ κάποιον κίνδυνο, γιατί ε, θα είναι επικίνδυνο να πω κάτι τέτοιο. Ε, λοιπόν, έχουμε σύστημα εμπορίας εκπομπών στην αεροπορία, αυτή είναι η αλήθεια θα πρέπει να μειωθούν οι δωρεάν άδειε. και επιπλέον για να υπάρξει κάποιο πλαφόν στις εκπομπές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Κόρσια το οποίο θα εγκριθεί νομίζω πολύ γρήγορα και βεβαίως η αντιστάθμιση των εκπομπών θα πρέπει το Κόρσια λοιπόν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν μπορώ να σα πω τώρα πώς. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να δούμε πώς θα εφαρμοστεί Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να δούμε πού πρέπει να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, ε, δηλαδή αφενός κάποια αναθεωρήση των κατευθυντηρίων γραμμών, απ' την άλλη να δούμε και το συνολικό δίκτυο και να δούμε αν κάποια τμήματα του μπορούν να γίνουν ε, κομμάτι του κεντρικού δικτύου. Αυτό αφορά βεβαίως ε, την αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ε, υπήρχε κάτι άλλο που αφορούσε τις ε, καθυστερήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν κομμάτι της ερώτησής σας. Έχετε πάλι τον λόγο κύριε Ζωτόσκη. Σας ε, ευχαριστώ. Τώρα δεν θέλω να σας αναγκάσω εγώ να συζητήσετε το πακέτο κινητικότητας, αλλά η δήλωση αυτή ότι θα αλλάξουμε τα όσα δεν λειτουργούν είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα υλοποιήσετε. Έχω άλλη μια ερώτηση τώρα. Μια ομάδα κρατών μελών ζήτησε να επεκταθεί το κύριο δίκτυο μέσω της Καρπαθίας Οδού. Αυτό είναι σημαντικό για την χώρα σας αλλά και για άλλες ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Γι' αυτό ακριβώς ε, κάνω την ερώτηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες ε, της Καρπαθίας Οδού. Δεν έχω κάποια απάντηση, λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να δούμε το βασικό δίκτυο, το συμπληρωματικό δίκτυο και να δούμε τι μπορεί να μεταφερθεί στο βασικό δίκτυο. Θα δούμε τις κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνουμε την εφαρμογή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών για να συμβούν αυτά τα οποία λέμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντέλη. Ο κύριος Ντέλη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Βάλιαν, είναι προφανές ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερη γραφειοκρατία για τι ε, επιχειρήσει των μεταφορέων. Στην επιστολή καθηκόντων της κυρίας Φοντερ Λάιεν σας ζητάει να εξασφαλίσετε ότι θα εφαρμοστούν πολιτικές που θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Τι μέτρα θα προτείνετε σε αυτή την πρώιμη φάση της εντολής σας, της θητείας σας, που θα μπορούσαν να μειώσουν το διοικητικό άχθος των επιχειρήσεων, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοιο. Κοιτάξτε, η προφανής απάντηση είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτομία για να εξυγχρονίσουμε το σύστημα. το σύστημα αλλά και σε ό,τι σημαίνει ως προς τους επιβάτες. Πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε εισιτήρια πολλαπλών συνδέσεων πρέπει να έχουμε συστήματα απεικόνησης των διαδρομών και των ανταποκρίσεων και πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό σύστημα που να είναι και ανθεκτικό έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τα δεδομένα που θα χρησιμοποιούμε σε συστήματα B2B. Και πάλι να είναι ασφαλή δηλαδή έναντι καταχρήσεων ή επιθέσεων του κυβερνού χώρου. η γραφειοκρατία στις μεταφορές είναι σε διάφορα επίπεδα. Σε κάποιες περιοχές έχουμε ψηφιοποίηση και εξυγχρονισμό. Έχουμε άλλες περιοχές, αλλά μέσα ίσως η σιδηρόδρομη να είναι το πιο προφανές, ή στα οποία διοικητικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται. Όμως η ψηφιακή τεχνολογία και ο συγχρονισμός συνολικά του συστήματος θα μείωνε τα διοικητικά εμπόδια που υφίστανται. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα νομοθετικών προτάσεων ή κανόνων που θα τροποποιούσατε, θα καταργούσατε, θα προτείνατε για να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα και επομένως την ε, δυνατότητα δημιουργίας θέσεων, νέων θέσεων εργασίας στις μεταφορικές επιχειρήσεις. Μιλάτε για την ανταγωνιστικότητα. Ο μιλητής είναι εκτός μικροφώνου. Δεν τον ακούν οι διερμηνείς. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Λέω θα κάνετε κάποιες τροποποιήσεις, θα προτείνετε κάποια καινούργια νομοθεσία ή ακύρωση παλαιότερων διατάξεων για να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα. Κοιτάξτε, ως Ευρωπαίοι πολιτικοί, λέει η κυρία Βαλέαν, γνωρίζουμε ότι η νομοθεσία πρέπει να ελέγχεται διαρκώς ως προς την αποτελεσματικότητα για την ανταγωνιστικότητα που έχει. Και όταν μιλούμε για έλεγχο κλιματικού αντικτύπου, πρέπει να μιλούμε και για έλεγχο ανταγωνιστικού αντικτύπου. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό επί της αρχής. Τώρα δεν θα μπορούσα να σας πω αν θα προχωρήσουμε σε πρόταση απόσυρσης του τάδε ή δίνα νομοθετήματος, θα πρέπει να αξιολογήσουμε συνολικά την επίδοσή τους ως προς την ανταγωνιστικότητα. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους επιτρόπους ως προς την αρχή του one in, one out και να έχουμε μια συνολική επανεξέταση της νομοθεσίας, λέει η κυρία Βάλεαν, και των συσχετισμών των νομοθετημάτων για τις μεταφορές με άλλους τομείς της οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί ε, κυρία Βάλεαν, ε, γνωρίζουμε τους στόχους του 2030, γνωρίζουμε τις δυσκολίες για τις επενδύσεις και τις ε, αδειοδοτήσεις. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε ένα καθεστώς προνομιακό. Έχω τρεις ερωτήσεις σε αυτό να σας θέσω. Ε, θεωρείτε ότι η προτεραιότητά θα πρέπει να εστιαστεί μόνο στο κεντρικό δίκτυο ή θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και το συνολικό δίκτυο. Επίσης ε, το θέμα της συντήρησης των υποδομών και του εξυγχρονισμού τους. στο ποσοστό που εμπίπτουν στα δημοσιονομικά μέσα. Επίσης, σχετικά με τη, μεταφορή του, με τη μεταφορά του Ταμείου Συνοχής για, προς τη διευκόλυνση για τις μεταφορές, αν και ε, τα ποσά που πρόκειται να μεταφερθούν δεν είναι ακριβώς, δεν συμφωνούν ακριβώς μεταξύ τους αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Κοιτάξτε, Core Network, το κεντρικό δίκτυο και το συμπληρωματικό δίκτυο. Πέραν των επενδύσεων στις ίδιες τις υποδομής έχουμε τις υποδομές με συγχωρείτε, έχουμε και τις επενδύσεις και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν υπάρχουν πάντοτε επαρκείς δυνατότητες ή ισότιμες δυνατότητες συντήρησης, μάλλον οικονομικής επιβίωσης των επιχειρήσεων συντήρησης για τον εξυγχρονισμό που χρειάζεται στις υποδομές, στα δίκτυα δηλαδή μεταφορών. Για τα πολυτροπικά μέσα, για τα ευφυή συστήματα κινητικότητας και τα λοιπά. Ως προς το βασικό και το συμπληρωματικό δίκτυο, για την ε, διευκόλυνση Connecting Europe, το μηχανισμό, πρέπει να διατηρήσουμε ένα καλό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο, αλλά ξεχνώ το τρίτο τμήμα της ερώτησής σας, λέει η κυρία Βάλεαν. 4 ή 11 δις ήταν από το Ταμείο Συνοχής. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχω την άποψη στη διαφορά, μεταξύ των επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου εδώ, η Τραν έχει δίκαιο και όχι η Ρέγγι, η Επιτροπή για τις Περιφέρειες, ως προς την κατανομή δηλαδή των κονδυλίων. Ο κύριος Ρικέ, συμπληρωματική, ευχαριστώ Πρόεδρε. Από τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή επίδοση, την περιβαλλοντική μάλλον επίδοση, πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ε, των υποδομών, του συστήματος, μέσω επενδύσεων κτλ. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και αποτρεπτική φορολόγηση. Για τα καύσιμα, για την κυροζήνη ή για τις εξωτερικές αναθέσεις των χερσαίων ταφορών. Αλλά το σχόλιο μου είναι η αύξηση εκπομπών, ε, είναι αύξηση όγκων και όταν έχουμε αύξηση όγκων των μεταφορών, δηλαδή των επιβατών, έχουμε και ένα θέμα δημοκρατικότητας των μεταφορών. Ε, γιατί όσοι δεν είναι στη θέση να πάρουν το αυτοκίνητό τους θα χρειαστούν μέσα συγκοινωνίας, μέσα μεταφοράς. Ε, και επομένως πώς μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα μέσο αποτρεπτικής φορολόγησης που θα επιβαρύνει τις τιμές. Επίσης ε, η οδηγία για τις για τις άδειε κυκλοφορίας, για τις ε, Eurovignette και οι διατάξεις της, ε, όπως και τα μέσα του προϋπολογισμού ε, σε σχέση με συγκεκριμένα κονδύλια σημαίνουν, πιστεύετε, επιταχύνεται, λέει η Πρόεδρος, ότι θα είναι δημοκρατικά αποδεκτοί αυτή οι φόροι εάν όντως βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των υποδομών και των μέσων. Και ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο για την ανοχή της. Κοιτάξτε, το εξωτερικό κόστος είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και λόγω της υφιστάμενης κατάστασης η αρχή οριπένων πληρώνει δεν εφαρμόζεται σωστά. Αν λάβουμε υπόψη μας το συνολικό όγκο χίλια δις. Και φορολογικά έσοδα 370 δις σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. ώστε να καλύπτουμε μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους μέσω του ρηπαίνοντος χρήστη. Δηλαδή ο ρηπαίνων χρήστη θα πρέπει να συνεισφέρει περισσότερα. Επομένως οι οδικές επιβαρύνσεις επί τη βάση της απόστασης και αυτό το λέει και η διάταξη του Eurovignette με μία πίστοση, με μία πρόβλεψη που είναι δύσκολη να την ποσοτικοποιήσουμε γιατί πολλά κράτη-μέλη, παρακαλώ ολοκληρώσετε λέει η Πρόεδρος, για την ελκυστικότητα των διατάξεων αυτών για το κοινό, ε, νομίζω ότι η αρχή ο, ο πληρώνει θα είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φουρόρε. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, για να συνδέσουμε καλύτερα την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρωθεί στους λεγόμενους ε, διαδρόμους, μεγάλες ε, σιδηροδρομικές αρτηρίες, οι οποίες συνδέουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό όμως δημιουργεί δύο προβλήματα, θεωρώ. Πρώτον, ε, οι μικρές κοινότητες είναι απομονωμένες και θα πρέπει άρα να πάνε στις μεγάλες πόλεις με αυτοκίνητο. Ειδικά στην Νότια Ιταλία όπου έχουμε πάρα πολλέ τέτοιες περιοχές στις οποίες δεν φτάνει ο σιδηρόδρομος. Ε, η πόλη Παραδείγματος η οποία ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ε, το 2019. Λοιπόν, και έχουμε ένα σχεδόν μονοπόλιο στο οποίο, από το οποίο εξαρτώνται οι εργαζόμενοι για να πάνε καθημερινά στην δουλειά τους. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση του κόστου. Μιλάμε για ένα 44% παραπάνω που πληρώνουν για το τρένο. Κάτι το οποίο είναι ντροπή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αποτελεσματική σύνδεση στην Ευρώπη, ειδικά στι μειονεκτικέ περιοχέ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποφευθούν οι καταχρήσει τη αγορά. Οι πολίτε ε, λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να δεχτούν κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ τιμές για να είναι χαμηλές, ε, αυτό γίνεται μέσω του ανταγωνισμού. Χρειάζεται λοιπόν ανταγωνισμό στην αγορά. Για να είναι χαμηλές όπως είπαμε. Λοιπόν πρέπει να επιβάλλουμε την ομοθεσία περί ανταγωνισμού. Όπως είπα θεωρώ ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις ε, της αγοράς και υποχρεώσεις που δεν εφαρμόζονται σωστά. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα κάνω εγώ είναι να αξιολογήσω το τι γίνεται και το τι δεν εφαρμόζεται και να προσπαθήσω να επιβάλλω την εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυρίας Φοντερ Λάιν υπάρχει μια οδηγία περί Ευρωπαϊκού Βασικού Μισθού για να καταπολεμηθεί το μισθολογικό dumping που κάνουν κυρίως οι ανατολικές χώρες. Συμφωνείτε με αυτό. Θα βλέπατε θετικά την εφαρμογή του και στον ε, τομέα των οδικών μεταφορών παραδείγματο χάρη όπου πληρώνονται πολύ χαμηλού μισθού. και τέλος θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των απομονωμένων περιοχών του Νότου, όπου θα θέλαμε ακριβώς να προσθέσουμε τους διαδρόμους αυτούς που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το πακέτο της κινητικότητας που προτείνεται δεν απελευθερώνει περισσότερο τις οδικές μεταφορές, οπότε θα έλεγα ότι βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας. Και βεβαίω ε, ο θεμητός ανταγωνισμός προωθείται μέσω της ε, καταπολέμησης των εταιριών, γραμματοκιβατίων και τα λοιπά. Και της συμπερίληψης τέτοιων πραγμάτων στην νομοθεσία. Για το κοινωνικό ντάμπινγκ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε... Ε, όχι, το ίδιο πράγμα λέω. Πρέπει να ενισχυθεί ο θεμητός ανταγωνισμός ε, για να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και μιλήσατε και για κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ και περνάμε στον κύριο Πίτερ Βιτένοφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλεάν. Η οδική ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στις οδικές μεταφορές. Υπάρχουν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μου, όπου τα θύματα των τροχαίων είναι πάρα πολλά και δεν μειώνονται. Στην αρχή της δήλωσής σας είπατε ότι βασικός ε, στόχος είναι να μειωθούν ε, στο μισό τα θύματα. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε. Δεύτερον, πολλές ευρωπαϊκές ε, πόλεις επιβάλλουν διαφόρους περιορισμούς και φόρους μεταξύ των οποίων στα αυτοκίνητα diesel. Αυτό επηρεάζει και τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων πώς ε, σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση δεδομένου ότι δεν υπάρχει ε, ένα ενιαίο πλαίσιο για την πρόσβαση στα αστικά κέντρα. Και η δικιά μου η χώρα τα πάει πολύ άσχημα στην οδική ασφάλεια και όπως είπα στην αρχή ε, είναι απαράδεκτα υψηλός ο αριθμός νεκρών και τραυματιών στην Ευρώπη, αν και παραμένει η ασφαλέστερη περιοχή του κόσμου. Για την οδική ασφάλεια, νομίζω ότι έχουμε δεσμευτεί σε ένα όραμα ε, μηδενικών θανάτων το 2050. Υπάρχει μια στρατηγική που έχουμε και σκοπεύω να την προωθήσω για να μειωθούν ε, οι σοβαροί τραυματισμοί στο μισό μέχρι το 2030. Βεβαίω, μιλάμε και για συγκεκριμένε δράσει, αλλά μιλώντα για την οδική ασφάλεια, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τομεί συγκεκριμένοι όπου πρέπει να παρέμβουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Είναι οι υποδομέ, η συμπεριφορά των ανθρώπων και η κατάσταση του στόλου των οχημάτων. Οπότε πρέπει να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για να δούμε το θέμα της οδικής ασφάλειας επιπλέον. Μπορούμε αυτό να το δούμε και μέσω του εξυγχρονισμού των έξυπνων συστημάτων μετάδοσης που θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η οδική ασφαλεία. Α, ναι. Για τους περιορισμούς η ποιότητα του αέρα στις πόλεις, η συμφόρηση, οι εκπομπές, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα δούμε με τρόπο ολοκληρωμένο. Οπότε έχουμε αυτήν την στρατηγική βιώσιμων μεταφορών στις πόλεις. Πρέπει να διευκολύνουμε την υιοθέτηση νέων τρόπων μεταφορών, μοιρασμένων, έξυπνων, της λεγόμενης ηλεκτρονικής κινητικότητας και της κινητικότητας ως, ως υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν θα συνεισφέρουν στην βελτίωση του αποτυπώματος των μεταφορών ε, στις ε, αστικές περιοχές. Βεβαίως υπάρχει επικουρικότητα, οπότε οι πόλεις ε, μπορούν να λάβουν τα δικά τους μέτρα και περιορισμούς. Αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για αυτήν την απάντηση. Ε, για τη δεύτερη μου ερώτηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ανατολική Ευρώπη είναι μια αγορά που έχει πλημμυρίσει δίζελ ε, από δεύτερο χέρι και ταυτόχρονα έχουμε περιορισμούς ε, στην κυκλοφορία τους. Χρειάζεται λοιπόν ένα γενικότερο πλαίσιο για την πρόσβαση οχημάτων ε, στις αστικές περιοχές. δεν μπορούν να θεωρηθούν πλέον τοπικά αυτά τα ζητήματα. Θεωρείται ότι χρειάζεται εναρμόνιση και ένα ενιαίο πλαίσιο. Νομίζω ότι έχουμε μια ήπια προσέγγιση. Κοιτάμε κατευθυντήρες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, το τι συμβαίνει στις αστικές περιοχές όπου περιορίζεται η πρόσβαση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι αναγκαίο για να λυθούν τα προβλήματα συμφόρησης και ποιότητας του αέρα. Θα προτιμούσα μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι τόσο κατακαιρματισμό, γιατί ο κατακαιρματισμός ε, εδώ είναι κακός ε, για όσους ε, ταξιδεύουν διασυνοριακά. Δηλαδή πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη και δεν ξέρουν το σύστημα που υπάρχει. Αυτό είναι εμπόδιο στην κινητικότητα. Απ' την άλλη αυτό πρέπει να το δούμε και με μεγαλύτερη διαφάνεια και πληροφορίες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοια μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ώστε να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Και θα δούμε αν απαιτείται περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μοντάρα. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, Αντίνα. Θα ήθελα να πω το εξή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ σήμερα το απόγευμα. Έχω κάποια ερωτήματα τώρα για τον ναυτιλιακό κλάδο. Μόλις τα αναφέρατε. Ο τομέας των ε, θαλάσσιων ε, μεταφορών με οδηγεί στην μπλε οικονομία. Η μπλε οικονομία ε, περιλαμβάνει δύο τομείς οι οποίοι είναι αναπόσπαστοι ε, μεταφορές και τουρισμός. Μιλάω για εμπορεύματα με τις υποδομές, ε, τουρισμό, κρουαζιέρες, μεταφορά επιβατών, όλα αυτά. Για να προωθήσουμε λοιπόν την πλέη οικονομία, θέλουμε μία επιτροπή και μία επίτροπο η οποία θα ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά. Τι είδου νομοθετικέ λοιπόν πρωτοβουλίε θα προωθήσει για την ευφύη ανάπτυξη στι θαλάσσιε μεταφορέ και πώ πιστεύεις ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να συντονιστούν με τον ωκεανό και το θέμα της δαλευμάτων. Ε, Απάντηση. Καταρχάς να πω ότι ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό είναι τμήμα της, επιτυχής, ε, της επιτυχίας μας. Αυτό που συμβαίνει όμως με τα υδατά ε, είναι προβληματικό. Αυτό το αντιμετώπισε και τμήμα του κανονισμού για την βιωσιμότητα, για τον αντικτυπο. Για το βιώσιμο αντικτυπό των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα και στα υδατά. Αν σκεφτούμε τι γίνεται με τη ρήπανση, με τα πλαστικά, τα πράγματα είναι τραγικά. Έχουμε όμως σχέδια για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη μεταφορά λιμάτων προς τους λιμένες. Αυτό είναι τμήμα των όσων προβλέπει η οδηγία, γιατί θεωρώ ότι και οι λιμένες και τα πλοία θα πρέπει να συμβάλλουν για το θετικό τελικά αποτύπωμα στα υδατά οι λιμένες ε, με την ε, συλλογή απορριμμάτων. Έχουμε νέες ιδέες σε ό,τι αφορά την συλλογή των απορριμμάτων αυτών από τα πλοία και από άλλους ε, ρηπαντές και από την άλλη θα πρέπει να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο τι γίνεται με τα πλοία και πώς συμπεριφέρονται όταν είναι στη θάλασσα. θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση να εφαρμοστούν οι πολιτικές και να μην καταλήξουμε να πετάμε στη θάλασσα αλευτικό εξοπλισμό και άλλα πολύ επιβλαβή στοιχεία. Ο τουρισμός συνδέεται άμεσα με τις μεταφορές. Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς μεταφορές. Και νομίζω ότι οι μεταφορέ συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ στενή λοιπόν αυτή η σύνδεση και από την πλευρά, πλευρά αυτή. Λυπάμαι που δεν είχατε θετική απάντηση, δεν είχατε απάντηση από την επιστολή που αποστήλατε στην ε, πρόεδρο Φοντερ Λάιεν. Δεσμεύομαι όμως να αγωνιστώ για να υπάρξει αποτέλεσμα από αυτή την άποψη. Η διευκρινιστική ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σα. Ένα δεύτερο σχόλιο και μία ακόμα ερώτηση. Τι μέτρα θα πάρετε ως προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων προς τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τη διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης στο Connecting Europe Facility. Υπάρχουν ε, καθυστερήσεις, υπάρχουν και κενά και προφανώς. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα κενά αυτά, ιδιαίτερα στις απόμακρες περιοχές. Εγώ είμαι από μία τέτοια περιοχή όπως τα γνωρίζετε. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, μιλάμε για αυξημένο κόστος, γεωγραφικά προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία ε, μπορεί να βοηθήσει το Connecting Europe Facility. Πώς θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν καλύτερα το CEF. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές απειλές. Έχουμε τόσες καθυστερήσεις. Αυτό προφανώς φοβίζει και τους ιδιωτικούς επενδυτές και είναι πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις καλές χρηματοοικονομικές ροές για τα προγράμματά μας. Υπάρχουν σοφείς αιτίε σε όλα τα έργα σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους, ε, τις δημόσιες συμβάσεις, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ήδη προτείναμε νομοθεσία, κανονισμό ή οδηγία για να μπορέσει να υπάρξει μια εναρμόνιση στις διαδικασίες αυτές. Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Και προφανώς θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά, να συντομιλήσουμε και με όλα τα κρατημέλη, γιατί για παράδειγμα η πρόταση να υπάρξει μία αρχή για να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα αυτά. Κάποια κρατημέλη διατείνονται ότι αυτό θα προσθέσει ένα επίπεδο γραφειοκρατίας. Αυτό δεν το θέλουμε προφανώς. και για να υπάρξουν πιο σύντομε περίοδοι διετή, για παράδειγμα, για την υλοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταλή. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Μιλάτε για την βιώσιμη α, κινητικότητα και την α, περιβαλλοντική ουδετερότητα. Αυτό σε ό,τι αφορά την αεροπορία. Μήπως μας πάει σε διαφορετική κατεύθυνση, λέτε. Φαίνεται λες και κρύβεστε πίσω από αυτό το πρόγραμμα για τους, ε, τον Single Sky, ενιαίο ουρανό, ε, λες και είναι κάτι μαγικό. Μιλάτε για στόχους για μείωση των εκπομπών, αλλά έχετε αποκλείσει τη χρήση φορολογία για την επιτεύξη αυτού του στόχου. Είπατε ότι θα το εξετάσατε αυτό. Δεν έχετε υπόψη ότι το εξετάζει αυτό η Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου έτους ε, αναφέρει τι θα σήμαινε η αύξηση της φορολογίας χωρίς να υπάρξει αντικτύπωση ε, στο εισόδημα. Λέτε ότι προωθείτε το σιδεροδρόμο. Πώς προωθείτε το σιδεροδρόμο όταν ουσιαστικά επιδοτείτε την αεροπορία, δεν υπάρχει φόρος ε, για τα καύσιμα, δεν υπάρχουν άλλοι φόροι. Γιατί υπάρχουν δηλαδή πτήσεις μεταξύ Βρυξελών και Άμστερνταμ. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι στα τρένα. Θα ήθελα να απαντήσετε τις ερωτήσεις που σας κάναμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για αυτή την ε, αγώνα προς τα κάτω. Δεν ε, έχετε... Δεν, έχετε, δεν είσαστε ενήμεροι για το γεγονό ότι πολλέ αεροπορικέ εταιρείε χρησιμοποιούν ψεύτικε ψευδοσυμβάσει. Κοιτάξτε, όχι, δεν κρύβομαι πίσω από τίποτα. Δεν έδωσα πιο πολλέ λεπτομέρειε γιατί ξέρω ότι τα ξέρετε αυτά. Και τα ξέρετε καλύτερα και από μένα τι γίνεται με όλες αυτές τις πρακτικές που δεν είναι καλές πρακτικές και προφανώς θα πρέπει να επιληθούν και προς την κατεύθυνση αυτή δεσμεύομαι γιατί χρειαζόμαστε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον για την ε, αεροπορία προκειμένου να συνεχίσει να είναι επιτυχής και επικερδής ως κλάδος. Για τις εκπομπές θα το πω ξανά και το επαναλαμβάνω ως σημείο αρχής θεωρώ ότι ο φόρος αυτός είναι τμήμα της λύσης μόνο. Δεν λέω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει φορολογία. Αν θέλετε να δεσμευτώ και να πω ότι δεν πρόκειται να αποκλείσει το ενδεχομενο φορολογησει φορολογήση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είπα ήδη ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ήδη εφαρμόζουν φόρο Ζήνης. Και λειτουργεί καλά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το συζητήσαμε αυτό με το Σώμα των Επιτρόπων, γιατί προφανώς αυτό είναι σοβαρή απόφαση. Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της ε, αεροπορίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την ε, ανταγωνιστικότητα του κλάδου στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ξέρω κάποιοι θα ήθελαν και θα προτιμούσαν η αεροπορία στον, στη φάση αυτή να μην υποστηρίζονταν και να έμπαινε ως πρώτη στην προτεραιότητα ο σιδηρόδρομος. Το καταλαβαίνω αυτό και δεσμεύομαι ότι θα επικεντρωθώ στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου με χαμηλότερε τιμές, γιατί όντω δεν χρειάζεται να πάρουμε μία πτήση από τις Βρυξέλλες στο Άμστερνταμ, αλλά τον θα δείτε τη τιμή του εισιτηρίου του τρένου, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι φτηνά και τα τρένα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς με ένα συνδυασμό μέτρων μπορούμε να πετύχουμε τέτοιους, ε, τέτοια μείωση της χρήσης της αεροπορία. Επίσης, αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση των καυσίμων. Αυτό συζητάω στο Single European Sky, γιατί χρειάζεται να υπάρξει εξοικονόμηση καυσίμων και αποτελεσματική χρήση των καυσίμων. Να δούμε λοιπόν τι τεχνολογικές τι τεχνολογικά επιτεύγματα υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή στο θέμα της φορολογίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιτάπητος, δεν κρύβομαι πίσω από τίποτε και δεσμεύομαι να τα εξετάσω όλα αυτά και να τα χρησιμοποιήσω για να μειωθούν οι εκπομπές στην αεροπορία και να καταστούν οι σιδηρόδρομοι πιο ελκυστικός τρόπος μεταφοράς και για επιβάτες αλλά και για αγαθά. Αυτό δεν απαντάει την ερώτηση. Είπατε ότι δεν θα εξαιρέσετε την φορολογία. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να λέτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει φορολογία για να αλλάξει η πολιτική στον τομέα αυτό. Έχουμε επιστημονικά α, τεκμήρια που το, που το τεκμηριώνουν αυτό. Ξέρω ότι αναφέρετε ότι θα κάνετε αναθεώρηση της ε, τη κεντρική νομοθεσία για την ενέργεια. Αυτό θα πάρει όμω τουλάχιστον πέντε χρόνια, γιατί χρειάζεται ομοφωνία. Και υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη που αντιτάσσονται. Ω Επίτροπο, θα είσαστε ηγετικοί σε ό,τι αφορά πολυμερείς και ε, διμερείς στον τομέα αυτό, γιατί αυτό χρειάζεται για το κλίμα. Και αυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει. Και το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί δεν μιλάμε μόνο για του εργαζόμενου. μιλάμε για την ασφάλεια επίση στην αεροπορία, το οποίο έχει βασικό ρόλο αν ε, λοιπόν συμφωνείτε με ένα προσωπικό το οποίο είναι κουρασμένο, κακοπληρωμένο και πετάει όταν δεν θα πρέπει να πετάει, προφανώ επηρεάζεται και η ασφάλεια του επιβάτη. Αυτό λοιπόν είναι. Και αυτό γίνεται όταν ε, του εκμεταλλεύονται οι αεροπορικέ επιχειρήσει. Δεν είναι ένα θέμα ανταγωνισμού αυτό. Η κυρία Βαλέαν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέω και πάλι είναι το εξής. Το είπα και προηγουμένω. Όταν κάποιο εισαγάγει ένα φόρο, υπάρχει το, ο κίνδυνο να αυξηθεί η τιμή. Το οποίο θα έχει φυσικά συνέπειε για την κινητικότητα του κόσμου. Ο κόσμο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφορά. Άρα, ο φόρος αποτυπώνεται σε κόστος κατά του καταναλωτή. Τα χρήματα αυτά πάνε στον εθνικό προπολογισμό γιατί δεν υπάρχει καμία αγγίηση απολύτως ότι αυτά τα χρήματα, αυτοί οι φόροι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθούν όλα αυτά που αναφέρατε, μείωση των εκπομπών, ε, οι συνθήκε εργασία των εργαζομένων του κλάδου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξετάσω. Αυτό λέω. Μιλάτε για τη δέσμευσή μου στον τομέα της αεροπορίας λες και δεν ξέρω ή λες και αδιαφορώ για τα θέματα αυτά. Δεν στέκει τίποτα από τα δύο. Εξοικειώνομαι με όλα αυτά τα θέματα. Τα οποία εσείς τα κατέχετε εδώ και καιρό, γιατί εργάζεστε εδώ και καιρό σε αυτά. Εγώ λοιπόν ενημερώνομαι για τα θέματα αυτά εδώ και δύο μέρες. Δεν θέλω λοιπόν να κρυφτώ πίσω από τίποτε, αλλά σκέφτηκα ότι αν δεσμευτώ για να συνεργαστώ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με το Κοινοβούλιο, για να επιλύσουμε τα προβλήματα και να βρούμε το σωστό τρόπο προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να μετακινείται με σωστές εύλογες τιμές, να υπάρχουν μέσα μεταφοράς ε, σωστά συμπεριλαμβανομένη της αεροπορίας, αυτό θα ήταν αρκετό. Αυτό από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιραντίνο, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ε, εισήγησή σας και τις απαντήσεις που δώσατε. Είναι αρκετά δύσκολο να παρεμβαίνει κανείς στο τέλος μετά από τόσες ερωτήσεις που έχουν ακουστεί. Αλλά πιστεύω ότι το ιδιαίτερο πεδίο με το οποίο θα ασχοληθείτε αξίζει να επαναλαμβάνουμε κάποια ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά εμπόδια ακόμα για τους επιβάτες στις μεταφορές. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Τα διάφορα σύστημα αγοράς των εισιτηρίων δεν είναι σύμβατα μεταξύ τους και δεν εξασφαλίζουν τα δικαιώματα του, επιβάτη ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί. Και αυτά πρέπει να αρθούν προκειμένου να έχουμε ένα λειτουργικό και ομοιογενές σύστημα το οποίο να διευκολύνει του επιβάτε. Αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι με προτέσεις εξίσου συγκεκριμένες και απτές. Πολλέ περιφερειακές περιοχές, ιδιαίτερα στον νότο της Ευρώπης, ενέχουν δυσκολίες που αποτρέπουν πιο οικολογικές επιλογέ που θα μπορούσαμε να έχουμε και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν, πρέπει να ε, ε, ολοκληρώσετε λέει η Πρόεδρος, Εμποδίζουν λοιπόν την επιλογή άλλων μέσων. Τι μπορείτε να κάνετε για να είναι πιο αποτελεσματικέ οι δημόσιε μεταφορικές υπηρεσίες. Κοιτάξτε, οι συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να υποστηριχθούν ως επιλογή για τους επιβάτες. Και πράγματι μερικά συστήματα αγοράς εισιτηρίων είναι, αποτελούν εμπόδιο ώστε να περάσει κανείς από το ένα μέσο στο άλλο. Χρειάζεται εδώ λοιπόν να εξυγχρονίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε μέσα νέας τεχνολογίας, νέες ψηφιακές λύσεις, να συνεργαστούμε με τους ενδιαφερομένους φορείς στο πεδίο αυτό, επί των δεδομένων και της χρήσης τους, της ακριβούς πληροφόρησης που πρέπει να έχει για τα δρομολόγια των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ άλλων, ώστε να μπορούν οι επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια πολυτροπικά και να είναι αξιόπιστα αυτά ως προς τα δρομολόγια που αναφέρουν. Όταν ένας επιβάτης αλλάζει μέσο μεταφοράς, αν έχει αγοράσει χωριστά το εισιτήριο για το κάθε μέσο, δεν είναι σαφές πώς καλύπτονται τα δικαιώματά του στη μία διαδρομή και στην άλλη. Πρέπει λοιπόν στις πολυτροπικές συνδέσεις να εξασφαλίσουμε όταν υπάρχει, όταν γίνεται η ανταπόκριση μεταξύ μέσων, να καλύπτονται τα δικαιώματα του επιβάτη. Γιατί ένα πράγμα είναι να χρησιμοποιήσει ένα λεωφορείο και ένα άλλο πράγμα, λέει η κυρία Βάλα, είναι να χρησιμοποιείς ένα αεροπλάνο. Ένα λεπτό έχετε ακόμα στη διαθεσή σας, λέει η πρόεδρος, στον κύριο Φιραντίνο. Ευχαριστώ την κυρία Βάλεαν, αλλά σας θυμίζω ότι για να διευκολύνουμε τις επιβάτες και ώστε οι δημόσιες μεταφορές να είναι πιο ελκυστικές με ευεργετικές επιπτώσεις και για τον τουρισμό που είναι σημαντικότατος για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Νότου της Ευρώπης, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα για να ενσωματωθούν τα τεντή, τα δίκτυα των μεταφορών, που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα καλής λειτουργίας και καλής ανάπτυξης του τουρισμού. Δεν θεωρείται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συσχετίσει τις μεταφορές και τον τουρισμό σε ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Γύρια κυρία Είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τα έχει συνδυάσει αυτά είναι σε καλύτερη θέση να τα δει συνολικότερα, να τα εξετάσει συνολικότερα. Είναι προφανές και το αντιλαμβάνομαι ότι ο τουρισμός δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί χωρίς μεταφορές. Νομίζω ότι στη μελλοντική δουλειά της ομάδας της Επιτροπής θα πρέπει πολύ να δουλέψουμε στα θέματα μεταφορών και τουρισμού και συζητώντας αυτό το θέμα στο Κολέγιο των Επιτρόπων νομίζω ότι ε, τα δύο χαρτοφυλάκια θα μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε ώστε να τα εξετάζουμε από κοινού, λέει η κυρία Βάλλαν. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιούτα Πάουλους, για ένα λεπτό, είναι μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Καλώ ήλθατε στην Επιτροπή μας. Κυρία Πάουλους. Καλησπέρα. Χαίρομαι για το ότι είπατε ξεκάθαρα ότι οι εκπομπές ε, της ναυτιλίας θα μπουν, πρέπει να μπουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και γνωρίζετε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί υπάρχει ήδη μια αξιολόγηση αντικτύπου και εκεί πέρα έχουν εργαστεί με μια τιμή του ETS γύρω στην σημερινή οπότε δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν προτάσεις που δεν κάνουν διακριτική μεταχείριση των ευρωπαϊκών πλοίων. Θα αφορά δηλαδή όλα τα πλοία που δένουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια Κάτι το οποίο λοιπόν είναι φθηνό και εύκολο να ενσωματώσουν τις, ε, το κόστος του ETS ε, και να τις ε, μετακυλήσουν στους πελάτες. Και Βεβαίω, αυτό σημαίνει ότι θα απορροφηθούν ε, τα πιστοποιητικά εκπομπών που υπάρχουν ήδη, οπότε δεν ξέρουμε αν θα μειωθούν οι εκπομπέ. Ερώτηση. Εάν ο κύριος Τίμερμανς ε, το κάνει θα το στηρίξετε εσείς. αυτό το οποίο ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε είναι να περιληφθεί η ναυτιλία στο σύστημα ETS. Νομίζω ότι είναι δυνατόν και ότι έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία με την εισαγωγή του ETS σε άλλους κλάδους και γνωρίζω ότι πρέπει να γίνει σωστά και να λειτουργεί καλά για να έχουμε μια υψηλή τιμή άνθρακα, αλλιώς δεν έχει νόημα. είναι δουλειά του κυρίου Τίμερμαν ακόμα για να το προτάνει, ε, να το προτείνουμε στο πλαίσιο της κλιματικής δράσης για να δούμε το πώς θα λειτουργήσει ακριβώς, αλλά βεβαίως εξαρτάται από εμάς, ε, Επίτροπο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το ορίσουμε με έναν τρόπο ώστε ε, μην χρειάζεται παρέμβαση για να λειτουργήσει λόγω τιμής της, ε, των δικαιωμάτων. Οπότε σε αυτήν την φάση δεν μπορώ να ξέρω ποια μέτρα θα ληφθούν. Απλά σας λέω ότι ε, εγώ είμαι προσυλλομένη και θα έπρεπε να είστε κι εσείς για να εισαχθεί ένα τέτοιο μέσο για τις εκπομπές στην αυτιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Είπατε πως ε, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ε, στην επιστολή. Αναφέρονται επίσης ε, και τα εναλλακτικά καύσιμα ως μια δυνατότητα. Όμως το μόνο εναλλακτικό αυτή τη στιγμή είναι το LNG υγροποιημένο φυσικό αέριο. Με αυτό όμως δεν θα μειωθούν οι εκπομπές γιατί εξακολουθεί να είναι ορυκτό καύσιμο και δεύτερον πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εκπομπές ε, μεθανίου στην αλυσίδα αλλά και στο ίδιο το πλοίο ε, έχουν ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στο θερμοκήπιο και δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Οπότε γιατί αναφέρεται αυτό το καύσιμο και όχι καύσιμα χωρίς άνθρακα για να προωθήσουμε την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πλοίων. Ακούστε, ναι. Ναυτιλία. Μάλιστα. Είναι πρόκληση για μένα το θέμα. Είχα κάποια πορεία σε άλλους κλάδους, αλλά εδώ πέρα μαθαίνω. της αρχής θα έλεγα ότι πρέπει να τα δούμε όλα και να ενθαρρύνουμε και μέτρα αγοράς ε, ανάπτυξη πιο βιωσιμών καυσίμων. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι στην αυτιλία δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει και δεν υπάρχουν και τόσο πολλές ε, λύσεις. Αλλά γνωρίζουμε τις εξελίξεις. Και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς, ε, αυτές τις λύσεις που είναι πιο βιώσιμες αυτή τη στιγμή και να ενθαρρύνουμε νέες ε, τεχνολογικές εξελίξεις, νέα ερευνητικά προγράμματα για να προχωρήσουμε ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερα το LNG γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι εύχριστο και υπάρχουν βιώσιμα βιοκαύσιμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το βασικό είναι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μου αρέσει επίσης ε, η ιδέα του πράσινου πλοίου. Θα μπορούμε να το δούμε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει και τα καύσιμα και άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι ώστε το πλοίο του μέλλοντος να είναι θωρακισμένος προς το κλίμα. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Έτιεν. Ε, κυρία Βαλεάν. Εδώ πάω πίσω σας είμαι. Να αναφερθώ στα θέματα του νέου ευρωπαϊκού ουρανού που ανέφερε ο Χωσέραμον ήδη. Α, θα μπω εγώ σε λεπτομέρειες. Έχουμε τώρα την δυνατότητα να επιτύχουμε κάποιους εύκολους στόχους με το ΣΕΖΑΡ. Συμφωνείτε ή θεωρείτε να, ότι είναι καλύτερη η πρόταση της Επιτροπής Σοφών. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, θεωρείτε ότι βρέπει, θα πρέπει να θέσει πρώτη τους όρους πριν από τη ΣΥΠΑ. Τρίτη ερώτηση για τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών. Κάποιοι τα προτείνουν και για τρένα και για πλοία. Ποια είναι η άποψή σας. Θα ήταν θετικό να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κυρία Βαλεάν. Η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. πρέπει να προσπαθήσω πίσω να εγκριθούν αυτά. Και ελπίζω οι πολιτικές εξελίξεις να μας φέρουν εκεί να επιτύχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Τι άλλο είπατε, τα μη επανδρομένα μάλιστα χαιρετίζω το ότι έχουμε ήδη ένα πλαίσιο ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πως θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε είμαι υπέρ μιας αγοράς για αυτές τις ε, ε, συσκευές, αλλά χωρίς όρους, με όρους ασφαλείας ε, και αποτελέσει τμήμα της νέας κινητικότητας ειδικά σε αστικές ε, περιοχές, ε, υπηρεσίες. Θα δούμε λοιπόν τι προϊόντα θα μπουν στην αγορά και θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την αγορά. Γιατί έχουμε νέες ιδέες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα αρκεί να είναι ασφαλή για τα στοιχεία των επιβατών. Αυτό συνδέεται με την ασφάλεια των μεταφορών Έχουμε τη συμφωνία με ΙΠΑ και Καναδά. Νομίζω πάει καλά, θα αξιολογηθεί. Δεν θα έλεγα ότι είμαι υπέρ για το σιδηρόδρομο, γιατί πολύ απλά νομίζω ότι οι ανάγκες του κλάδου είναι τελείως διαφορετικές. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους <coughs> και να δραστηριοποιηθούμε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε τρένα. Αλλιώς ο κόσμος δεν θα τα εμπιστεύεται. Και αυτό πρέπει να στηρίξουμε το τρένο. Ε, έτσι ακόμη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαλεάνα. Σε ό,τι αφορά το Single European Sky έχουμε μια πολύ ανοιχτή πρόταση του 2014. Είναι παλιά η πρόταση αυτή. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση. Προτιμάτε να βολευτείτε με τις εύκολες λύσεις μία ενιαία και σύντομη διαδικασία για την εφαρμογή όλων των τεχνικών προτύπων σε ό,τι αφορά την κοινοπραξία. Ή προτιμάτε να ακολουθήσετε τις προτάσεις του Αντιπροέδρου για να συλλέξετε πιο πολλέ απόψει για το πώ θα πρέπει να λειτουργήσει το Single European Sky και για τα ανεπάντατα οχήματα δεσμεύεστε να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα για τη νέα νομοθεσία για τα ανεπάντατα οχήματα. Απάντηση. Ναι, τώρα κατάλαβα λίγο καλύτερα την ερώτησή σα για το Single European Sky. Νομίζω ότι προτιμάω να πετύχω αυτά που μπορούμε να πετύχουμε τώρα γιατί χρειάζεται εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Και νομίζω ότι χάνουμε χρόνο. Έχουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δεν έχει και νόημα, δεν λειτουργεί το σύστημα όσο έχει τώρα. Και μετά να, να το σκεφτούμε όσο θέλουμε και όσο χρειάζεται για τα ανεπάνδρωτα οχήματα. Φαντάζεστε ότι τέτοιου είδου λεπτομέρειε εσεί τη γνωρίζετε και εγώ δεν τη γνωρίζω, αλλά είναι θέμα αρχή ότι θέλω να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι είναι θετικό να γίνει. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο και τελευταίο. Στον κατάλογο ο κύριο ε, Μαριάν Μαρινέσκο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλεάν, για τι απαντήσει σα. Είπατε δικαίως και σωστά ότι η κοινωνική πτυχή είναι πολύ σημαντική για όλους τους τρόπους μεταφορών και προφανώς και για την αεροπορία. Η ΆΖΑ, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Ασφάλεια στην Αεροπορία, έλαβε ευθύνες και προς την κατεύθυνση αυτή στον κοινωνικό κλάδο. Συνεργάζεστε με την ΕΑΖΑ για να εισαγάγεται κανόνες σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση στη δευτερο... δευτερογενή νομοθεσία σε ό,τι αφορά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης. Κύριε Μαρνέσκο, δεν είμαι εμπειρογνώμων και δήμων σε θέματα αεροπορίας όπως είστε εσείς και διάφοροι άλλοι συναδελφοί και όντως εισαγάγονται οι κοινωνικές πτυχές και ναι θα συνεργαζόμουν με την ΕΑΣΑ για να μπορέσω να εισάγουμε να αγαγούμε στην νομοθεσία και την κοινωνική πτυχή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Μαρνέσκου. Δεύτερη ερώτηση για τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα είναι πάντα πολύ σημαντικά. Μπορούμε να δεσμευόμαστε για ό,τι θέλουμε στις μεταφορές, αλλά ούτε η Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε τα καρδιμέλη θα μπορούσαν να πετύχουν τίποτα χωρίς ε, χρηματοδότηση. Είχαμε δυσάρεστες εμπειρίες πριν από πέντε χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιέκοψε στη σοφία του τον ε, γενικό προϋπολογισμό και η πιο μεγάλη περικοπή που έγινε, έγινε στο ΣΥΕΦ. όπως το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Θα χρησιμοποιήσετε όλοι σας την αρμοδιότητα και την εξουσία ως μέλος ε, της Επιτροπής για να μην υπάρξουν περικοπές άλλα στο ΣΕΦ και αν θα υποστηρίξετε κατά δεύτερον την ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για ένα ποσό 4 δισεκατομμυρίων όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντηση. Νομίζω ότι όλοι οι επίτροποι θέλουν να υπερασπιστούν τον προπολογισμό τους, αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το CEF είχα αναστατωθεί ιδιαίτερα όταν το Συμβούλιο περιέκοψε τον φάκελο για το ΣΕΦ e στον τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύω όμως ότι στο μεταξύ τα καλά αποτελέσματα στο πλαίσιο του ΣΕΦ e απο... τα αποδέχονται όλα τα κράτη-μέλη και έχει αποδείξει την αξία του και την επιτυχία του το πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι την φορά αυτή οι πόροι για το ΣΕΦ δεν θα βρουν αντίθετο το Συμβούλιο. Πώς θα προσπιστώ τώρα την ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, γιατί φυσικά χρειαζόμαστε πιο πολλά χρήματα σε πάρα πολλά προγράμματα. Και ιδιαίτερα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τις βιώσιμες και φύσεις μεταφορές, χρειαζόμαστε ό,τι πόρους διαθετούμε και επίσης να διατηρήσουμε και τους πόρους στα Ταμεία Συνοχής και για την στρατιωτική κινητικότητα. Έχουμε και τον ορίζοντα 2020 και υπάρχουν ακόμα πόροι στον ορίζοντα Ευρώπη και αυτά τα χρήματα επίσης τα χρειαζόμαστε για τον εξυγχρονισμό του συστήματος και σε ό,τι αφορά το InvestEU θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τους πόρους αυτούς στο έπακρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την ακροματική διαδικασία, τις ερωτήσεις. Ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, αλλά και για το γεγονό ότι τηρήσατε το χρονικό όριο και καλώ την κυρία Βάλεαν να κάνει μια σύντομη δήλωση αν θέλει ολοκλήρωσης. Επιθυμείτε κυρία Βάλεαν. Παρακαλώ. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Αγαπητή Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι, που είχατε την υπομονή να με ακούσετε σήμερα. Από όλα τα ερωτήματά σας, από όλες τις παρατηρήσεις, αυτό που συγκρατώ πάνω απ' όλα είναι ότι ο τομέας των μεταφορών είναι μια οικογένεια ανθρώπων που έχουν διάφορα ενδιαφέροντα αλλά που επιθυμούν να εργαστούν μαζί για μια περιοχή μεταφορών πιο ευφυή, πιο αποτελεσματική, πιο συμπεριληπτική, με καλύτερες συνθήκες εργασίας για αυτούς που εργάζονται και για αυτούς που χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα. Εγώ δεσμεύομαι για τους στόχους αυτούς, αλλά με όλες σας τις ε, ερωτήσεις αντιλαμβάνομαι την περιπλοκότητα και τις πολλές και διάφορες ανάγκες που έχουμε να καλύψουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, πρέπει να κινητοποιήσουμε πόρους και πρέπει να είμαστε ευφυείς στην προσέγγιση μας. και να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Εγώ επαναλαμβάνω ότι τοποθετώ τους ιδιοδρόμους στο κέντρο της προσπάθειάς μου, αλλά χρειαζόμαστε κάθε έξυπνη ιδέα, κάθε ευέλικτο και ευφυές μέσο, ώστε να προαγάγουμε τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, Πρέπει να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους σε όλα τα μέσα μεταφορίας τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών και αυτά που προσπαθούσα να σας πω καθ' όλη τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας είναι ότι εσείς είστε οι δήμονες στο θέμα αυτό. Στο συγγνώμη αν οι απαντήσεις μου δεν ήταν επαρκώς εξειδικευμένες, αλλά έχετε τέτοιο βάθο λεπτομέρειες διαθεσή που εγώ δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να σα υποσχεθώ είναι ότι πολύ σύντομα θα ξέρω πολύ περισσότερα. Και είμαι σίγουροι ότι θα συνεργαστούμε για να βρούμε λύσεις για τις ανάγκες του συστήματος. ευχαριστώ και πάλι που είχατε την υπομονή να με ακούσετε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ευχαριστούμε την κυρία Βάλεαν. Ολοκληρώνεται εδώ η ακροασία. Ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι, ε, αγαπητά μέλη. Ευχαριστούμε την κυρία Βάλεαν, ευχαριστούμε για τις γραπτές απαντήσεις που μας αποστήλατε προς την Επιτροπή Τραν. Για τους ε, δημοσιογράφους θα έχουμε συνέντευξη τύπου σε λίγα λεπτά, στις 4 υπάρχει χρόνος, στον δεύτερο όροφο, μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και θυμίζω στους συντονιστές και αντιπροέδρους ότι η συνεδρίαση αξιολόγησης θα λάβει χώρα 4 και μισή και κλεισμένων των θυρών. Ολοκληρώσαμε εδώ, σας ευχαριστώ.